Äh, Κυρίες και κύριοι, κυρίσω την έναρξη συνεδρίασης. Είναι καθοδόν ο κύριος Βάρον που θα έρθει σε λίγα λεπτά. Να πούμε μερικά διαδικαστικά όμως προηγουμένως. Μία παράκληση έχω. Από τις 3 και 4 θα με αντικαταστήσει εδώ στο Προεδρείο ο κύριος Ταγιάννη, διότι από τις 3.30 και μετά υποδέχομαι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κολομβίας. Ε, Ήταν ε, κάτι, μια ανηλυμένη υποχρέωση που υπήρχε πριν εγγραφεί ε, η ημερησία διάταξη, στην ημερησία διάταξη διάσκεψη των Προέδρων. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να ματαιώσω το ραντεβού μαζί του και θα αναλάβει ο κύριος Σταγιάννη να προεδρεύσει από τις 3 και 4 εδώ. Σας ερωτώ λοιπόν, έχετε ιδιαίτερες επιθυμίες, αν όχι. Μέχρι να έρθει ο κύριος Παρόμπαι να εκμεταλλευτούμε το χρόνο και να τον αξιοποιήσουμε, όχι. Όλοι είστε ευτυχείς και χαρούμενοι, χωρίς καμία επιθυμία. Ωραία. Διακόπτω και πάλι μέχρι να έρθει ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Έχω κάποια επιθυμία, αλλά δεν μπορείτε να υλοποιήσετε και όλες μας τις επιθυμίες. Ναι, όντως. Έχετε απόλυτο δίκιο αν κάτι ισχύει είναι αυτό ακριβώς. Ε, μακάρι να μπορούσα να ικανοποιήσω όλες τις επιθυμίες. Κανένας δεν υποχρεώται στα αδύνατα. Καλώ Καλώς. Καλώς ορίσατε θερμά κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή τη μικρή καθυστέρηση και οι δύο πρόεδροι ε, πήγαν ε, από το πρωτόκολλό μας στη συνεδρίαση ε, της Επιτροπής Υγείας δεν ξέρω που είναι σε άλλο κτίριο. Ανησυχούσαν για την υγεία τους και τους πήγανε στην Επιτροπή Υγείας. Δεν ξέρω τι να πω. Σας ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος του Κοινοβουλίου για την καθυστέρηση αυτή. Εμείς φταίμε. Κυρίε και κύριοι, πριν κηρύξω την έναξη συνεδρίαση και δώσω το λόγο στον κύριο Βαρόμπεϊ, επιτρέψτε μου μία σύντομη παρατήρηση ως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι είναι η τελευταία δημόσια διάσκεψη των Προέδρων που παρίσταται ο κύριος Φανρόμπόη ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ε, παρουσιάζει την ενημέρωση για την τελευταία συνεδρία του Συμβουλίου. Κύριε Φανρόμπόη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το έπραξα και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά να το επαναλάβω και εδώ επιθυμώ ενώπιον των συναδέλφων αυτό που είπα εκεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Φρονώ ότι με το αξίωμα που αναλάβατε πριν από πέντε έτη, που ήταν ε, αχαρτογράφητα ύδατα, αναλάβατε μία από τις πιο δύσκολες αποστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι μας γνωρίζουμε τους 28 κυρίες και κυρίους ε, που είναι υπό την δική σας προεδρία με διαφορετικό χαρακτήρα. Με ισχυρό, εγωιστικό ή μη ε, και πρώτα απ' όλα εκπροσωπούν τα συμφέροντα των κρατών τους. Με κειμενόμενη αυτοπεποίθηση. Είναι Ηράκλειος ο άθλος που αναλογεί στον πρόεδρο ε, και που θα πρέπει να έχει κανείς την ηρεμία σας, την ισορροπία σας ε, και την ε, σαφήνεια και την αποφασιστικότητα για να καταλήγετε σε συμβιβασμούς. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε επιφυλάξεις ε, για τη δημιουργία καν του Προέδρου του Συμβουλίου και αμφιζητούσαν την ίδια την ύπαρξη. Εσείς πραγματικά ήσασταν εξαιρετικός ε, ήμουν και εγώ από τους επικριτές, είδα όμως ε, και είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω το πώς εργάζεστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με ευγνώμων για την προθυμία πάντα για συνεργασία αλλά και το σεβασμό τον οποίο επιφυλάξατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είμαστε πάντα σύμφωνοι με ε, τον προγραμματισμό των Συμβουλίων, γιατί τις περισσότερες φορές συνέπιπταν με τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούμε την επόμενη περίοδο <laughs> να το αλλάξουμε αυτό, αλλά δεν έχει σχέση αυτό ούτε με την ποιότητα της δικής σας δουλειάς, ούτε άλλαξαν ε, καθόλου ούτε επηρέασαν την ποιότητα της συνεργασίας μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω κύριε Ρόμπαϊ στην τελευταία αυτή συνεδρίαση για τη συνεργασία, ε, αλλά και πολύ προσωπικά το Χέρμαν και να ευχηθώ ότι καλύτερο για το μέλλον. Στο τέλος, στις ε, φωτογραφίες, είχαμε δύο οικογενειακές φωτογραφίες. Είχαμε μία την ε, γνωστή, τη θεσμική, με τους πρωθυπουργούς, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και τους θεσμικούς, που είναι η κανονική οικογενειακή φωτογραφία και μετά μια πραγματική οικογενειακή φωτογραφία. Ο κύριος Φαρόν με τα παιδιά του, τους γαμπρούς και τις νύφες του και τα εγγόνια του. Ήταν από τα πιο συγκινητικά αυτά που ζήσαμε και όλα τα παιδιά ήταν φρόνημα. Μόλις έφτασε ο Κάμερον άρχισε το πιο μικρό να κλαίει. Δεν ξέρω, νομίζω τυχαίο θα ήταν αυτό μάλλον. Ε, ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή αυτή και είμαστε ευγνώμονες ε, όλοι ε, που είχαμε την ευκαιρία να τη ζήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και ό,τι επιθυμείτε για το μέλλον. Mr. President. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, καταρχήν Μάρτιν, σε ευχαριστώ θερμά για τα ευγενικά σου λόγια με ιδιαίτερη χαρά θα σα ενημερώσω για τη διάσκεψη κορυφή του Οκτωβρίου, το τελευταίο σύνοδο κορυφή ε, από τη δική μου Προεδρία. Και θα το κάνω με το γνωστό μου ύφο και στυλ. Δεν πρόκειται να αλλάξω γιατί είναι τελευταία φορά. Ήταν αξιομνημόνευτη η Σύνοδο Κορυφή, όχι γιατί επιτύχαμε συμφωνία για την ενέργεια και το κλίμα στην Ευρώπη ε, για το 2020-2030, αλλά γιατί μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις ανθρωπότητας ε, και μία για την οποία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίστηκε. Το Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε θέσει ως καταληκτική προθεσμία τον Οκτώβριο και τήρησε την υπόσχεσή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προσφέραμε σταθερότητα στους οικονομικούς τελεστές για να μπορέσουν να προγραμματίσουν τις επενδύσεις τους, ε, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και να περάσουμε σε ένα πιο βιώσιμο πλανήτη, να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, στους απογόνους μας. Και μάλιστα το ειδικό πάνελ για το κλίμα εξέδωσε την έκθεση που ζήτησε δραστική μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου για να σταματήσουν οι κλιματικές αλλαγές. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, η υλοποίηση μέχρι το 2030 μείωση ως 40% που είναι από τους πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους στον κόσμο. Με την απόφαση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταβιβάσει ένα πολύ θετικό μήνυμα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Ένα αισιόδοξο κλίμα και κλίμα με, και, ε, ε, δε, πολύ φιλόδοξε δεσμεύσει. Βέβαια, μερικέ χώρε μέλη θα επιθυμούσαμε περισσότερε φιλοδοξίε στον ένα ή στον άλλο τομέα. Αλλά μην υποτιμάτε τη σημασία της υλοποίησης της σύναψης αυτής της συμφωνίας και μάλιστα ένα χρόνο πριν από την διάσκεψη κορυφής των Παρισίων για το κλίμα, το Δεκέμβριο του 2015. Τώρα θα είμαστε σημείο αναφοράς ε, για τις επόμενες διαπραγματεύσεις ε, για το περιβάλλον. Και μετά την συμφωνία, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕΟ ο Μπαν Κιμούν, χαιρέτησε την Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που συνεχίζει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον κόσμο και είπε ότι οι κλιματικές, οι στόχοι θα πρέπει να γίνουν ε, σημείο αναφοράς ε, και στη συζήτηση στι Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα έχουμε τέσσερις στόχους ε, εμβληματικού που ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση. Θέλουμε πιο φιλοπεριβαλλοντική ενέργεια, πιο ασφαλή και λιγότερο δαπανηρή. Καταρχήν, αποφασίσαμε εγχώρια μείωση τουλάχιστον 40% των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030. Και μάλιστα τα σημεία αναφοράς για το 1990 είναι δεσμευτικά. Και έχουμε φιλόδοξους, πολύ φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους για το 2050. Ε, οι περισσότερες προσπάθειες θα γίνουν από το σύστημα εμπορίας εκπομπών στους τομείς ενέργειας και βιομηχανίας. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την παγκόσμια μας ανταγωνιστικότητα και θα πρέπει να παρεμποδίσουμε την βιομηχανία μας με τις φιλοδοξίες μας. Φυσικά έχουμε και τους τομείς που είναι εκτός ε, συστήματος εμπορίας εκπομπών και θέλουμε εθνικούς τους στόχους ώστε να γίνουν συλλογικές προσπάθειές μας όσο πιο αποδοτικές γίνονται. Επίσης, καθαρή ενέργεια. Ε, είπαμε τουλάχιστον 27% μέχρι το 2030 είναι το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και μάλιστα ο στόχος αυτός είναι δεσμευτικός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και στον τομέα αυτό η τεχνολογία ε, προχωράει ακάθεκτη και ραγδαία. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει και η νοοτροπία μας και ως προς αυτό κάποιες λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν αργότερα. Αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή ενέργεια το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι γύρω στο 14%. Οπότε 27% και παραπάνω μέχρι το 2030 μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει τουλάχιστον να διπλασιάσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι οι καθαρές πηγές ενέργειας. Τώρα, ενεργειακή ασφάλεια. Είπαμε να αυξηθεί κατά 20% ε, και η ενεργειακή απόδοση. Είναι ενδεικτικό αυτό το νούμερο όμως σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα και σε σχέση με τις προβλέψεις για το 2030 με την τρέχουσα κατανάλωση και τεχνολογία θα γίνει μια αναθεώρηση το 2020 και για το 2030 θέλουμε ε, νέο επίπεδο, 30%. Θέλουμε να μειώσουμε επίσης την ενεργειακή μας εξάρτηση ένα άλλο ζήτημα ιδιαίτερα φιλές σε όλους. Γνωρίζω ότι στο Κοινοβούλιο έχετε σημαντικές απόψεις υπέρ της ενεργειακής απόδοσης και, έχουμε, και θα έχετε τη δυνατότητα να διατρανώσετε τη θέση σας από τη στιγμή που θα υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις. Τώρα, διασυνδέσεις ενεργειακές για να διαχειριστούμε την προσφορά και ζήτηση διασυνοριακά και επίσης ε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της μείωσης της εγχώριας ενέργειας. Μέχρι στη... Θέλουμε 15% διασυνδεσιμότητα μέχρι το 2030 και να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα προγράμματα διευρωπαϊκά ώστε να ελοποιήσουμε τους στόχους μας και στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο. Συγκεκριμένα προγράμματα θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσουμε απλές διακηρύξεις ε, και να δημιουργήσουμε μια πραγματική ενεργειακή ένωση. Ένα όραμα και σχέδιο που ε, είναι ιδιαίτερα προσφυλές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συζητήσαμε επίσης και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Η οικονομική ανάκαμψη είναι πιο αργή από ό,τι ελπίζαν πολλοί. Και μετά την επαναφορά της σταθερότητας στην Ευρωζώνη τον, ε, το φθινόπωρο του 2014. Βέβαια, χαμηλή ανάκαμψη οφείλεται στη μείωση του δυναμικού ανάκαμψης που αυτή τη στιγμή είναι σήμερα 0,05% ο αριθμός ανάκαμψης. Και αυτό οφείλεται στην υψηλή ανεργία και στο χαμηλό επίπεδο επενδύσεων. Θαύματα δεν υπάρχουν. Η ανάπτυξη είναι το άθροισμα της αύξησης των ορών εργασίας και της ανταγωνιστικότητας. Η έλλειψη επασχόληση, η έλλειψη θέσεων ε, εργασίας και η έλλειψη των επενδύσεων δημιουργούν τεράστιες πιέσεις. Ε, γι' αυτό ε, πολύ, προσπάθεια συγκυριακής ανάπτυξης προσκρούει στα διαρθρωτικά μας προβλήματα. Επίσης έχουμε γεωπολιτική αστάθεια που διαβρώνει την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και οι επιδόσεις των χωρών BRICS είναι ε, χαμηλότερες από ό,τι περιμέναμε και για την Κίνα και για τη Βραζιλία και τη Ρωσία και αυτές οι ε, χαμηλές επιδόσεις επηρέασαν τις εξαγωγές μας και την σχετική ανάπτυξη των χωρών της Ευρωζώνης που έχουν εξαγωγές προς χώρες αυτές η νομισματική μας πολιτική είναι θετική. Δεν συνέβαλε στην έλλειψη της οικονομικής ανάπτυξης. Τώρα έχουμε και τη δημοσιονομική πολιτική. Ούτε και αυτή επηρέασε αρνητικά την ανάπτυξη το 2014. Τα τελευταία χρόνια επιδείξαμε ευελιξία στη δημοσιονομική μας πολιτική. Δίνοντας έμφαση όχι στο ονομαστικό έλλειμμα, αλλά στο διαρθρωτικό έλλειμμα. Και οι επιπλέον προθεσμίες που δόθηκαν το 2013 για να ε, βρεθούμε κάτω από το 3% σε σχέση με το, τη συνθήκη της, ε, του Μάστριχτ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τώρα, ως προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία των αγορών εργασίας, να καταπολεμήσουμε τις αντιπαραθέσεις μεταξύ αυτών που είναι εντός και εκτός, μεταξύ αυτών που είναι προνομίχοι και προστατευμένοι και εκείνων που έχουν επισφαλείς θέσεις εργασίας, ε, που είναι νέοι, μετανάστες, γυναίκες. Επίσης θέλουμε μια αγορά, την ψηφιακή αγορά, την ενεργειακή ένωση και φυσικά μια πραγματική ζώνη έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτησε τι προθέσει τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει 300 δισεκατομμύρια ενάυσματα για τις επενδύσεις ε, τα επόμενα χρόνια. Έτσι θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να κάνουν πιο μεγάλε επενδύσεις ε, και η τόνος των επενδύσεων προϋποθέτει δράσεις και στην προσφορά αλλά και στη ζήτηση. Η παρούσα οικονομική κατάσταση είναι περίπλοκη, γιατί έχουμε όχι μόνο ασθενείς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και εξαιρετικά χαμηλό πληθωρισμό. Και μάλιστα αυτό ισχύει περισσότερο στις χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό φυσικά βαρύνει την κατάσταση και στη, δημόσιο χρέος και στο, στο ιδιωτικό χρέος. Ήδη η χρέωση είναι υπερβολική και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Θα πρέπει λοιπόν ε, χωρίς ταμπού, χωρίς φόβους, χωρίς έμονες ιδέες και χωρίς ιδεολογίες να κινητοποιήσουμε κονδύλια έχοντας και βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους με σεβασμό των ε, ιδρυτικών αξιών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Γιατί όλο μας το σύστημα στηρίζεται στην ανάπτυξη και την απασχόληση έχουμε επίγνωση της κατάστασης αυτής. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, της Ευρωζώνης ζήτησε από τους τέσσερις προέδρους ε, μία έκθεση το Δεκέμβριο για, την, ε, για τον ενισχυμένο οικονομικό συντονισμό. Απαραίτητο βήμα κατά τη γνώμη μου για να υλοποιήσουμε μία γνήσια, μία θετική οικονομική και νομισματική ένωση. Μία άγουσα που χαράξαμε και στην προηγούμενη έκθεση του 2012. Ε, αγαπητοί βουλευτέ, και τι εξωτερικέ υποθέσει συζητήσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μιλήσαμε για τη μάστιγα του έμπολα στη Δυτική Αφρική. Αλλά χάρη στι σοβαρέ δεσμεύσει άμεσα και κατά τη διάρκεια τη συνάντηση για ένα δι ευρώ που θα αφιερωθεί στην καταπολέμηση του ιού έμπολα, θα πρέπει απλώ να φροντίσουμε να ε, χρησιμοποιηθεί σωστά το ποσό αυτό. Ε, συντονισμός επίσης θα αναλυθεί από τον Επίτροπο Στυλιανίδη που θα αναλάβει τα καθήκοντά του για τα θέματα αυτά. Συζητήθηκε λοιπόν όπως έγινε σε, όλα τα, σε όλες μας τις συναντήσεις από το Μάρτιο και θα συνεχίσουμε να συζητούμε το θέμα αυτό και στο μέλλον για τις σχέσεις μας για την Ουκρανία και θα ζητώντας από την ε, Ομοσπονδία της ε, Ρωσίας να αναλάβει τις δεσμεύσεις της βάσει της συμφωνίας του Μίνσκ. Αναμένεται ο χειμώνα και η τροποποίηση λογοδοσία μας στο αέριο, αλλά και αντιδράσεις στις εκλογέ στην Ουκρανία ήταν πολύ αρνητικές ως τώρα. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, ήταν το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό στο οποίο προέδρασα. Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι ε, πάντοτε έδρασα και κινήθηκα στο όνομα του ευρωπαϊκού συμφέροντος. Αυτό δεν το λέω ως κάτι αφηρημένο, αλλά το ευρωπαϊκό συμφέρον είναι, είναι το σύνολο, το άθροισμα 28 εθνικών συμφερόντων. Ε, και ήταν και ένα επίτευγμα να φτάσουμε στους 28 για να συμφωνήσουμε κάθε φορά με τον καθένα ξεχωριστά γύρω από ένα τραπέζι διπραγματεύσεων. Όχι πάντοτε ε, διαμιάς και πολλές φορές με πάρα πολλή ε, προσπάθεια για ανταλλάγματα και διαπραγματεύσεις. Αλλά AUTHORWAVE καταφέραμε να αποδείξουμε ότι το αδύνατο μπορεί να λειτουργήσει, ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ενιαία ως 28 κράτη-μέλη. Ελπίζω ότι η επόμενη πενταετία θα, είναι, ε, θα δώσει εξίσου θετικά αποτελέσματα στους κρίσιμους καιρούς που περνάμε, όπως και η προηγούμενη πενταετία. Χρειαζόμαστε θέσεις απασχόλησης για να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων. Τα τελευταία πέντε χρόνια είδαμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να συνεργαστούν και είμαι γι' αυτό ε, ευγνώμων στον προηγούμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε αγαστά από την ε, πρώτη ημέρα μέχρι τη συνεργασία μας μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Χάρη στην σταθερή παρουσία του Ευρωκοινοβουλίου, με το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον Προέδρο του Μπούζεκ και Σούλτ, ε, όλα πήγαν καλά. Επίση, πολλέ επαφέ είχα διαρκώ και με πολλού και πολλές από εσάς. Βεβαίως κάποιες φορές έχουμε διαφωνίες και διαφορά στις ε, απόψεις μας. Όμως δεν έχουμε ανταγωνιστικό ρόλο ως θεσμικά όργανα. Εξυπηρετούμε τον ίδιο σκοπό, τον ευρωπαϊκό σκοπό, δηλαδή την ευημερία όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζω αυτό ε, καθορίζει το έργο των ε, θεσμικών μας οργάνων, το οποίο τα οποία είναι το ίδιο εκτεθειμένα στην κοινή γνώμη και εμείς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εσείς στο Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δώσω τώρα ε, το λόγο για πρώτη φορά επισήμως ε, στον κύριο Γιούνκερ, νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αξιότιμε κύριε πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κύριε πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι. Δεν απευθύνομαι σε εσά για πρώτη φορά. Έχω την εντύπωση ότι ε, πολλές φορές χρειάστηκε εδώ να μιλήσω μετά από δική σας πρόκληση. Με χαρά λοιπόν θα έρθω να σας εξηγήσω ε, σε λεπτομέρειες το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχει συγκληθεί γι' αυτό η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Σε μερικές εβδομάδες θα μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Ε, είναι η τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου που μας απασχολεί σήμερα, που είχα την ευκαιρία να ε, συμμετέχω. Αυτό είναι ένα ίδιο ε, της Ευρώπη. Συμμετείχα σε τέσσερα ευρωπαϊκά συμβούλια, χωρί να είμαι καν πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Είχε την καλοσύνη πάντα μου να με προσκαλεί ο κύριο Φαν Ρόμπαϊ για να ακούω τι απασχολεί τι κυβερνήσει. γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να τι γνωρίσω αυτέ τι κυβερνήσει. Βέβαια, έχω συμμετάσχει σε πάνω από 120 συμβούλια ευρωπαϊκά στη ζωή μου, οπότε δεν ήταν και τεράστιε οι εκπλήξεις που έζησα εκεί, ήταν μάλλον σπάνιε. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, σε σχέση με την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή κτλ. Διότι δεν ήμουν ενεχόμενο μέρος εκεί στις διαπραγματεύσεις και στις συζητήσεις, παρόλο που ενστερνίζομαι απολύτως τα συμπεράσματα που ε, εξήχθησαν. Ανέθησα στον αρμόδιο αντιπρόεδρο που έχει τα ενεργειακά θέματα να ε, μεταφέρει στην πράξη τώρα όλα αυτά τα συμπεράσματα ε, του Συμβουλίου. Θα σας παρακαλέσω να προσκαλέσετε στις συνεδριάσεις σας που λέτε ότι είναι δημόσιες και τον Αντιπρόεδρο Σεύσκοβιτς για να σας ενημερώσει ε, ως προς τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες, τις προτάσεις, τις προθέσεις, ακόμα και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, θα ζητήσω από τον Επίτροπο Άρης Κανιέτε που ε, έχει στο χαρτοφυλάκιό του την ενεργειακή και την κλιματική πολιτική να κάνει ό,τι μπορεί, έτσι ώστε το Δεκέμβριο του 2015 στη διάσκεψη των Παρισίων να είναι στη θέση Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάσει μια συμπαγή και συντεταγμένη θέση σχετικά. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα στη συζήτηση του Συμβουλίου για θέματα οικονομικά και ιδιαίτερα στο Συμβούλιο του Ευρωζώνης ε, που προείδρευσε ο Χέρμαν Φάρομπαϊ για τις πρωτοβουλίες. Χαίρομαι πάρα πολύ που και ε, τα δύο αυτά συμβούλια ενέκριναν επί της αρχής το επενδυτικό πρόγραμμα που θα αφορά 300 δισεκατομμύρια και σας είχα εξαγγείλει κατά τη διάρκεια της ε, ομιλίας μου στις 15 Ιουλίου επί τη αναλήψη των καθηκόντων μου και προτίθεμαι να παρουσιάσω το πρόγραμμα αυτό πριν τις ε, διακοπές των Χριστουγέννων. Μην νομίζετε ότι επειδή είμαι Άγιος Βασίλης θα το κάνω αυτό, αλλά επειδή πιστεύω ότι είναι πήγοντα τα θέματα. Δεν θα ήθελα ακόμα σήμερα να μπω σε λεπτομέρειες. Για το επενδυτικό πρόγραμμα θα προεδρεύσω αύριο στην πρώτη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αύριο το πρωί, όπου θα αρχίσουμε αυτή τη σημαντική εργασία που είχα αρχίσει ήδη από τον Αύγουστο, χωρίς να μου έχει δοθεί εντολή, αλλά δεν είμαι ακόμα σε σημείο ούτε σε θέση, ε, χωρίς τη συμφωνία του Σώματος των Επιτρόπων, να σας ανακοινώσω διάφορες ε, προθέσεις που αφορούν κυρίως τον ιδιωτικό τομέα και όχι τόσο το δημόσιο. Γιατί δεν έχει έρθει η ώρα να αυξηθεί το δημόσιο χρέο και τα ελλείμματα στην Ευρώπη. Αν αυξηθεί το δημόσιο χρέος και για να υπάρξει αϊφόρος και μόνιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη η προϋπόθεση είναι τα ελλείμματα, θα έπρεπε να είχαμε ήδη ξέφρενη ανάπτυξη, πράγμα που δεν ισχύει. Άρα ε, θα πρέπει να συνδυάζονται οι πολιτικές εξυγίανσης των προϋπολογισμών που είναι εκ των όνου κάνευ με τις ε, ανατολισμένες προς την απασχόληση και την εργασία πολιτικές. Με χαρά ε, είδα να μου ανατίθεται η Προεδρία των Προέδρων που θα προβληματιστούν για την καλύτερη διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη και ε, υπό την προεδρία ήδη του κυρίου Φαν και ως πρόεδρος του Eurogroup είχα την ευκαιρία και την τύχη να ε, συμμετάσχω στην εκπόνηση μιας έκθεσης των τεσσάρων προέδρων πριν από δύο χρόνια και τώρα συνεχίζω αυτή την προσπάθεια ως πρόεδρος των τεσσάρων πρόεδρων και με το Δεκέμβριο να παρουσιάσω τα κυριότερα στοιχεία ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε αυτό το νοδικό χάρτη προς μια καλύτερη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης που αξίζει να βελτιωθεί διότι σε πολλές περιπτώσεις χωλαίνει ακόμα και αν έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι. Well, Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δεν θα σχολιάσω τα θέματα ούτε της ενέργειας ούτε των εξωτερικών, γιατί ο πρόεδρος Φανρόμπαη το έπραξε. Θα συνεργαστώ όσο γίνεται πιο στενά με τον Κοινοβούλιο και στο παρελθόν. Επί δεκαετίες έχω έρθει ως υπουργό Εργασίας, Οικονομίας, Οικονομικών, Πρωθυπουργό, κάθε φορά στο Κοινοβούλιο ερχόμουν. Και θα με βλέπετε όποτε με καλείτε ή ακόμα και όταν δεν θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, το λόγο έχει ο Βέμπερ, πρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φανρόμπαη, διότι ε, μετά από δική μας απόφαση ε, αποφάσισε και το Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρχισε να εργάζεται ε, ο κύριος Γιούνκερ με τους Ευρωπαίους επιτρόπους και χρονικά συμπίπτηκε πολύ καλά η σημερινή συνεδρίαση με την αυριανή της Κομισιόν. Το βασικό θέμα, ενέργεια και κλίμα. Θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω από πλευρά του ΕΛΚ αυτά που είπε ο κύριος Φωνρόμποη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα ε, και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε ότι είμαστε φιλόδοξοι στους στόχους μας ως Ευρωπαίοι. Είναι σημαντικό αυτό. Η Ευρώπη είναι παγκοσμίω υπόδειγμα για τη συμπεριφορά ε, ως προς το κλίμα και την ενέργεια και για το μέλλον και ελπίζω αυτό το μήνυμα να πιάσει τόπο και στο Παρίσι και παγκοσμίως. Ελπίζουμε ε, στο Παρίσι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για δεσμευτικό στόχο και όχι για προαιρετικούς και ε, μη δεσμευτικούς. Πιστεύουμε ότι το 40% δεν είναι κάτι που πρέπει να υποτιμούμε. Αν καταλάβουμε ότι από το 1990 μέχρι σήμερα έχουμε εξοικονομήσει ε, όσο θέλουμε να εξοικονομήσουμε τα επόμενα 10 χρόνια, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ό,τι εξοικονομήσαμε σε 20 χρόνια, τώρα το έχουμε ως στόχο για 10 χρόνια. Είναι φιλόδοξος ο στόχος και δεν θα πρέπει η Ευρώπη ίδια να υποτιμά τον εαυτό της. Και θα ήθελα να πω επίσης από πλευρά του ΕΛΚ ότι ε, με όλες τις συζητήσεις που κάνουμε θα πρέπει πάντα να έχουμε ε, ρεαλιστικούς στόχους. Βεβαίως να προχωρούμε στεναρά, αλλά να μην τρέχουμε και χάνουμε τους στόχους μας. Η πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια συνδέεται και με τις τιμές της ενέργειας. Γι' αυτό η αδυναμία στην ανάπτυξη στην Ευρώπη ε, και τα κλιματικά ζητήματα θα πρέπει να ε, συνυπολογίζονται. Για την μείωση θα ήθελα να πω το εξή ακόμα. Τα προβλήματα που έχουμε για τους στόχους μείωσης έρχονται την ε, εφαρμογή του στην πράξη. Ωραία η στόχη, αλλά όταν αρχίζουμε να μιλάμε για καφετιέρες ή για λαμπτήρες πυρακτώσεως στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε που πάνε οι συζητήσεις και δεν καταλήγουν θετικά για την Ευρώπη ε, στα μάτια του κόσμου. Γι' αυτό θα πρέπει, Ζαν Jean-Claude Juncker, μαζί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί πώς θα επιφέρουμε και μια ισορροπία θα πρέπει τα κράτη-μέλη όταν λαμβάνονται αποφάσεις για την ενεργειακή απόδοση, ας πούμε, για την εφαρμογή στην πράξη, να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να μην προσπαθούν να ξεγλιστρούν ότι α, δεν ξέρω τίποτα αυτή η απόφαση λήφθη στις Στα ενεργειακά δίκτυα έχει γίνει κάποια πρόοδος, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ε, περιοχές ε, για να προχωρούμε. Πρέπει να γίνει επιτέλους αυτό να υλοποιηθεί και ελπίζω να προχωρήσουμε και για την εσωτερική αγορά σίγουρα θα είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πολύ κατακερπαντισμένο δίκτυο και διανομή. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Γενικά για την ενεργειακή πολιτική δυστυχώς στο Συμβούλιο υπάρχει και ένα θέμα διαδικαστικό. Δηλαδή ε, όταν έχουν ε, κάποια επίπτωση στη βιομηχανία αποφάσεις θα πρέπει να διατηρείται ομοφωνία. Το είπε και ο πρόεδρός μας στη συνεδρίαση αυτή, ότι αυτό δεν συνάδει απολύτως αυτή τη στιγμή με τις συνθήκες. Ε, το Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις επί της αρχής για το μέλλον, κάνει προτάσεις ή κομισιόν και εκείνο που αποφασίζει είναι το Κοινοβούλιο. Ε, θέλω να υποστηρίξω αυτό που είπε ο Σούλτ ε, στην συνεδρίαση αυτή του Συμβουλίου, ότι κατά την άποψή μα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να τηρεί τις συνθήκες και από αυτού. Να μπω και σε κάποια άλλα θέματα που δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη, δύο, που ανησύχησαν όμως τη συζήτηση. Αυτά που είπε ο Ντέιβιτ Κάμερον για τους λογαριασμούς που καλείται να καταβάλει. Τώρα δεν του αρμόζει ε, αυτό ένα, σαν μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έναν εξέχοντα πολιτικό να είναι έξαλλος και να κοκκινίζει πούμε, και να παραφέρεται. Όταν συμφωνούμε στην Ευρώπη για κάποια θέματα, ε, δεσμεύεται και η Μεγάλη Βρετανία από τις συζητήσεις και τις συμφωνίες. Το δεύτερο που επίσης δεν ήταν στη μέση διάταξη, αλλά ανησύχησε, ήταν η συμπεριφορά του κυρίου Ρέντζη μετά από ε, μια επιστολή για τον προϋπολογισμό του και είπε δεν θα μου πούν οι γραφειοκράτες των Βρυξελών πώς θα κάνω τον προϋπολογισμό μου. Ε, τα λέω αυτά τα δύο γιατί κύριε Φανρόμποη σήμερα ε, παρευρίσκεστε ως απερχόμενος πρόεδρος και σας ρωτώ. Στο Συμβούλιο τα συζητάτε αυτά τα θέματα συμπεριφοράς και στάσεις Γιατί το θεωρώ απαράδεκτο. Αυτοί οι συνάδελφοι παίρνουν τις αποφάσεις από κοινού ή εν πάση περιπτώσει προκάτοχή του, κυβερνήσεις και μετά βγαίνουν και κάνουν τέτοιες απαράδεκτες δηλώσει για αποφάσεις των Βρυξελών υποτιθέμενες τι οποίες έχουν συμμετάσχει αυτοί. Να πούν οι άλλοι οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί, μα τι είναι αυτά που λες, συμφωνεί με αυτά που λέμε εδώ ή όχι. Ίσως τώρα στο τέλος της θητείας σας μπορείτε να μας πείτε αν τα συζητάτε αυτά με το όνομά του τα πράγματα και είναι, ή απλώς επιδεικνύεται κάποια ανοχή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές. Και ε, για την ανάπτυξη υποστηρίζω τα όσα είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής δεν είναι τα στοιχεία αυτά που θα επιθυμούσαμε, αυτά που χθε δημοσιεύτηκαν και θα παρακαλούσα τα κράτη-μέλη να υποστηρίξει το Jean-Claude Juncker ε, στο πακέτο το επενδυτικό και τέλος εξ ονόματος του ΕΛΚ ε, εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να εκφράσω τι ευχαριστήσεις ε, προσωπικά. Δεν είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ πολύ μαζί του γιατί είμαι νέος πρόεδρος. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Χέρμαν Βαν Ρομπέι. Άφησε τη σφραγίδα του. Ήταν μια νέα θέση που δημιουργήθηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας και όχι μόνο με, τη, με το ύφο του και με τον τρόπο του και με τη συμπεριφορά του. Και πραγματικά μπράβο σας που έχετε ε, αυτή την εικόνα, αυτή τη συμπεριφορά σας ταιριάζει και ταιριάζει και στο Συμβούλιο. Ο μάνατζερ, ο σοβαρός, ο διαμεσολαβητής μεταξύ διαφόρων συμφερόντων και ιστορικά, αν το κοιτάξει κανείς, ε, μπορεί να διαπιστώσει πόσο πολύτιμο είναι να έχουμε στην Ευρώπη ένα τέτοιο όργανο όπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντώνται ε, συχνά και διαπληκτίζονται και εναντιώνονται αλλά τελικά συμφωνούν και είναι πραγματικά μια ιστορική επιτυχία για την Ευρώπη που έχουμε αυτό το όργανο και με τη δική σας ηγεσία βεβαίως βελτιώθηκε πολύ. Θα ήθελα επίση να πω ότι στην κρίση ιδιαίτερα ήταν επίμαχο το θέμα της διακυβερνητικής συνεργασίας αλλά παρόλα αυτά απαραίτητο. Και εσείς είχατε πάντα ε, το βλέμμα σας στραμμένο προς τα πάνω, προς τις συνθήκες, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και κατά τη διάρκεια της κρίσης ε, ε, απαιτήθηκε δράση και ήσασταν δίκαιος διαπραγματευτής και στα θεσμικά ζητήματα και θα ήθελα να ευχαριστήσω ως πρόεδρος του ΕΛΚ, τον πρόεδρο του Συμβουλίου που προέρχεται από το ΕΛΚ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήσασταν ένας πολύ καλός μηχανοδηγός αυτής της ατμομηχανής ε, του Συμβουλίου. Στον επόμενο σιδηροδρομικό σταθμό θα κατεβείτε και θα ανέβει ο νέος μηχανοδηγός, ο κύριος Τούσκ. Σας ευχόμαστε ό,τι επιθυμείτε για το επόμενο διάστημα. Στη ζωή σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βέμπα. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Πιτέλα. Από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε Σούλτς. Θα συμφωνήσω και εγώ στα λόγια ευχαριστειών και ευγνωμοσύνης που εκφράσατε προς τον πρόεδρο Φαναμοπόη. Δεν ήταν απλό το καθήκον που ανέλαβε, ε, ήταν και κάτι καινούριο και ε, ήταν μεγάλη ευθύνη που έφερε σε πέρα ο μεγάλο κύρος και ιδιαίτερο στυλ ο κύριος Φαναμοπόη. Ευχαριστούμε λοιπόν. Νομίζω ότι σωστά ε, αναφερθήκαμε στις δηλώσεις του Συμβουλίου που για λόγους πολλές φορές και στατικικής γίνονται κατά τη διάρκεια μιας συνόδου και ε, σε σχέση με τα τελικά αποτελέσματα. Είδαμε ότι δεν μπορεί να κρίνεται η συμπεριφορά ενός ε, Πρωθυπουργού, του Πρωθυπουργού της Ιταλίας, κατά αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής και συνεπής οι δεσμεύσεις της ε, Ιταλίας έναντι της ε, Ευρώπης. Δύο μεγάλα ζητήματα απασχόλησαν το Συμβούλιο. Η οικονομία, οι κλιματικές αλλαγές και η εξωτερική μας πολιτική. Μου άρεσε πολύ η ιδιαίτερη επισημότητα με την οποία ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ είπε στο Στρασβούργο ότι αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η ιδιαίτερη υψηλή σημασία ευκαιρία, το είπατε αυτό με ιδιαίτερη σοβαρότητα κύριε Γιούνκερ και συμφωνώ. Δεν θα έχει μέλλον η Ευρώπη αν αποτύχουμε για άλλη μια φορά. Και δεν μπορούμε να αποτύχουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες των 6 εκατομμυρίων επιπλέον ανέργων, τον κοινωνικό αποπλισμό, την ε, ε, ένδια, τους ε, μακροοικονομικές απαιτήσει και τις κοινωνικές αποκλήσεις μεταξύ των κρατομελών. Δεν μπορούμε να αποτύχουμε ξανά σε έναν κόσμο όπου πολλοί μας χρειάζονται. Γι' αυτό το πακέτο για την ανάπτυξη και σε σχέση με τις επενδύσεις θα έπρεπε όντως να καταφέρει να αντιστρέψει αυτή την τάση. Πρέπει αυτή η δέσμη μέτρων να γίνει αντιληπτή κατά τον ορθό τρόπο ώστε να επιφέρει την σωστή ισορροπία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πόρων με νέα δημοσιονομικά ε, μέτρα ελέγχου, με τον καταμερισμό των στόχων και το ρόλο του ε, Κοινοβουλίου, του δικού μας, του Ευρωκοινοβουλίου που θα πρέπει να συμμετάσχει στην όλη μελέτη θα πρέπει να δούμε το σύνολο των μεγάλων αλλαγών που επηρεάζουν μια σειρά από εθνικές πολιτικές. Χρειαζόμαστε μεγάλη δυνατότητα μεταρρυθμίσεων ε, στην Ευρώπη και στα εθνικά κράτη-μέλη, ώστε να εξηγιανθούν τα δημοσιονομικά των κρατών μελών και να ανακάμψει η οικονομία για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Με την οποιαδήποτε ε, ε, δυνατότητα ευελιξία στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εδώ αυτό είναι ζωτική σημασία και χρειάζεται για να πετύχει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω και την σοιαλιστική κατάσταση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Ε, ε, Σόρευση πληρωμών και, δυνα... και περίπτωση πραγματικού πλήγματο στην αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βασικό μα δυναμικό, οι φοιτητέ, οι ερευνητέ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσει, οι ε, κοινότητε, οι αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση, τι περιφέρειες και του δήμου. όλα αυτά μόνο από τον Ευρωπαϊκό Προλογισμό μπορεί να στηριχθούν με την κατάλληλη πολιτική οικονομική αύξηση και ανάπτυξη, σε μια κρίσιμη καμπή για τι περισσότερε από τι χώρε μα, πολλέ είναι αυτέ που αντιμετωπίζουν σοβαρά και κοινωνικά προβλήματα. Carta αυτό είναι λοιπόν ένα πρώτο σημείο και έπειτα για τις κλιματικές αλλαγές. Σε αντίθεση με τον συνάδελφο Βέμπερ, θεωρώ ότι η συμφωνία την οποία πετύχαμε είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Ε, σε περίπτωση μη συμφωνίας βεβαίως, ε, εάν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ε, θα περιμένουμε τις εξελίξεις και στην ερχόμενη Σούπερ Σύνοδο Κορυφή στο Παρίσι του χρόνου. Αλλά δεν θα πρέπει να χάσουμε και το ραντεβού αυτό του Δεκεμβρίου του 2015, όπου η διεθνή κοινότητα και ο κόσμο περιμένουν ακριβώ ε, την ανάληψη δεσμεύσεων για δεσμευτικού ε, στόχου συγκεκριμένα. χωρί δεσμευτικού στόχου, δεν θα μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε το φαινόμενο τη αναθερμάνσης του πλανήτη και την, τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τον περιορισμό της αύξησης θερμοκρασίας μόνο σε δύο βαθμούς. Πρέπει να προστατεύσουμε τους φυσικούς πόρους, να προλάβουμε νέους πολέμους για το, για το νερό και τα τρόφιμα και την ε, περαιτέρω ε, ε, φτώχεια των επιπλέον πληθυσμών. Επίση, για την εξωτερική πολιτική, η κυρία Μογκερίνη ε, ήδη έχει αναλάβει δράση για όσα συμβαίνουν στην Μπουρκίνα Φάσο αυτέ τι ημέρε. Είναι ένα ανθρωπιστικό και πολιτικό δράμα αυτό που συμβαίνει. Θα πρέπει να καταδικάσουμε την ανάληψη εξουσίας με τα όπλα και να στηρίξουμε τις θεμητές προτάσεις του λαού της Μπουργκίνα Φάσο, απαιτώντας τον σεβασμό των θεμελίων του δημοκρατικού οικοδομήματος. Η ομάδα μου καταδικάζει το πραξικόπημα και ζητά με επιμονή το να γίνουν σεβαστά τα ε, βασικά δικαιώματα των πολιτών, ώστε η μετάβαση να γίνει από τους ελεύθερους πολίτες βάσει του συντάγματος. Θα πρέπει να ε, μην γίνουν αποδεκτή, να μην γίνει αποδεκτή αυτή η προσπάθεια ανάληψης εξουσίας. Και ακόμη και στην Αφρική, Πρόεδρε, πρέπει να ε, περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις για να ξεπεράσουμε την κοντόφθαλμη προσέγγιση που εδώ και χρόνια μας έχει εμποδίσει την οργανική μας σχέση με τον πρώτο μας συνομιλητή, σύμμαχο και εταίρο, την Αφρικανική Ήπειρο, να βελτιώσουμε και να αναθερμάνουμε τη σχέση μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καμάλ από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, πω στον Πρόεδρο του Συμβουλίου ότι η ομάδα μου είναι υπέρ ε, των στόχων των κλιματικών και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2003. Και χαίρομαι γιατί δεν έχουμε νέου ε, συγκεκριμένου εθνικού στόχου για τη γενικό στόχο ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και τέτοιο θα δημιουργήσει προβλήματα στι επενδύσει σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Αλλά χαίρομαι στην έμφαση που δίνεται στο συλλογικό χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει η ανάληψη αυτών των δεσμεύσεων. Αντί όμως να είμαστε πολύ συγκαταβατικοί για το στόχο του 30 και 40% θα πρέπει να να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο ώστε και στο επόμενο Συμβούλιο για το Περιβάλλον στο Παρίσι το 2015 να πείσουμε τους εταίρους μας γιατί θα είναι άχρηστο να μειώνουμε εμείς τις εκπομπές μας ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Βραζιλία, Κίνα, Ρωσία δεν τις μειώνουν αντίστοιχα. Επίσης χαιρόμαστε για τις αναγγελίες και τις δεσμεύσει που αναλύθηκαν για το έμπολα. Θα πρέπει να λυθεί και αυτό το θέμα υπόψη. Τώρα, επανέρχομαι σε ένα θέμα που επισήμαναν οι προλαλήσαντες ε, ένα θέμα που δυστυχώς στιγμάτισε την, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τις τεχνικές προσαρμογές ε, στις εθνικές εισφορές στον, στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Εσείς είπατε μόνος σας ότι θέλετε μια πιο πολιτική επιτροπή. Θα πρέπει κάποιοι να είδαν λοιπόν ε, το πολιτικό χαρακτήρα και τον δυνητικό πολιτικό όλεθρο μιας τέτοιας κατάστασης. Όταν μιλώ στους ψηφοφόρους μου στο Ηνωμένο Βασίλειο και στους φίλους στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ολλανδία, νόμιζαν ότι μας κάνουν πλάκα. Μου είπαν οι Έλληνες συνάδελφοι, μετά πόσα περάσαμε τα τελευταία χρόνια, μετά τη λιτότητα που μας ταλάνισε. Ζητάτε, μας ζητάτε να δανειστούμε περισσότερα χρήματα για να πληρώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πάνε στην ε, Γερμανία. Βλέπετε το πολιτικό χαρακτήρα αυτής της κατάστασης. Μου λένε οι Βρετανοί. Καθίστε μια στιγμή, είχαμε καλή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Μας τιμωρείτε γι' αυτό, ενώ μια χώρα όπως η Γαλλία ε, συνεχίζει να έχει ψηλά ελλείμματα. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η εντύπωση που έχουν οι πολίτες και αυτό είναι ο πολιτικός χαρακτήρας της κατάστασης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να αποφεύγουμε φράσεις ε, που λένε ότι οι υπολογιστές λένε όχι ή λένε περισσότερα ή είναι μόνο τεχνικές οι προσαρμογές. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα και σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί αύριο θα έχουμε την ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Ξέρουμε τι θα μας πει. Μπορούμε να λέμε ότι ε, οφείλεται αυτό στην ανευθυνότητα των κρατών μελών, αλλά δεν ακούν κάτι τέτοια οι ψηφοφόροι. Θα ρωτήσουν οι ψηφοφόροι γιατί δεν ανέλαβε τις ευθύνες της Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί δεν είχε σωστούς λογαριασμούς τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε αρμόδιο επίτροπο για τον προπολογισμό. Θα πρέπει να, να αναλύσουμε όλα αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να σταματούμε να να προσποιούμαστε ότι μειώνουμε τον προπολογισμό και ταυτόχρονα να ζητούμε συμπληρωματικέ εισφορέ από τα κράτη-μέλη. Και τέλο, κύριε Πρόεδρε, σα αναγνώρισαν ε, πολλοί ε, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, ω δίκαιο διαπραγματευτή και έντιμο διαμεσολαβητή. Και εμεί ω Ευρωβουλευτέ εκτιμήσαμε ιδιαίτερα τον τρόπο που χειριστήκατε τι επαφέ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και Νομίζω ότι η πολιτική σταδιοδρομία σας βοήθησε στην, τα τελευταία σας καθήκοντα. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία που είχαμε την τελευταία πενταετία και σας ευχόμαστε καλή τυχή για το μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Καμάλο, κύριο Φερχόφστατ από τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σήμερα είναι λίγο αλλαγή φρουράς η αίσθηση που δημιουργείται. Ο περχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βανόμπεϊ που Χαίρομαι, χαρά ε, τον συγχαίρω ε, για το έργο του και έχουμε και τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πολύ θα θέλαμε να συγχαρούμε και να χαιρετήσουμε για το έργο που θα έρθει και για τις προτάσεις του. Ξέρω ότι η συνεδρίαση αυτή έχει να κάνει κυρίως με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αλλά στον τύπο ειλικρινά δεν είδα πάρα πολλά άρθρα για την κλιματική αλλαγή. Τα περισσότερα άρθρα ήταν για ένα άλλο επεισόδιο που έκανε ο Κάμερον. Ο Κάμερον που από ό,τι φαίνεται έχει τώρα νέα στρατηγική είναι να κάνει επεισόδιο κρίση σε κάθε Ευρωπαϊκή Σύνοδο κορυφή. Αν γίνεται και κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβει ότι είναι κακή στρατηγική, γιατί ο κόσμος προτιμάει από το κακέκτυπο το αυθεντικό. Και η τελευταία κόπια της ιδέας του UKIP του κυρίου Κάμερον ήταν ενοχλητική και τελείως τρελή και για τους βασικούς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους Ευρωπαίους πολίτες και πρέπει να το το πούμε. Και πρέπει να πω, και είναι πολύ σπάνιο για μένα κύριε Καμάλ, ότι για αλλαγή συμφωνούμε με τον κύριο Κάμερον για την κρίση που προκάλεσε. Είναι κακό το σύστημα τεχνικές προσαρμογές στα τέλη του έτου, όπου πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στέλνει επιστολέ και να λέει ότι παίρνετε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κάποιοι άλλοι πρέπει να πληρώσετε περισσότερα στα τέλη του έτου. Αλλά όταν πει το α, μετά πρέπει να πει και το β. Γιατί ξέρουμε τι φταίει για το κακό σύστημα είναι ότι ο προπολογισμό της Ένωσης βασίζεται σε κρατικές συνεισφορέ και όχι σε γνήσιους ιδίου πόρου όπως είχε προβλεφθεί στην αρχική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδού ο λόγος. Οπότε, εάν ο κύριος Κάμερο θέλει πραγματικά να αλλάξει το σύστημα ε, των τεχνικών προσαρμογών αρκεί να ακολουθήσει ε, το αίτημα και την πρόσκληση και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής το συντομότερο να καθιερώσουμε ένα προϋπολογισμό και πολιετής προϋπολογισμούς που να βασίζεται στους ιδίους πόρους και στην άμεση χρηματοδότηση από τους πολίτες και όχι τεχνικές προσαρμογές σε κρατικές συνεισφορές. Και αυτό μου δίνει την ευκαιρία, Πρόεδρε, να μιλήσω λίγο για την αρχή της λειτουργίας της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρω ότι Κύριε Γιούνκερ, Ζαν έχετε νέα ιστοσελίδα. Α, ούτε, εσείς δεν το ξέρετε. Μάθετε το λοιπόν. Έχετε καινούργια ιστοσελίδα ε, και έχετε και ένα πολύ ωραίο λάβαρο στον πολύ χρωμό. Αυτό το έχετε δει. Α, ξέρετε τι γράφει. Μια νέα αρχή για την Ευρώπη. Ε, Αυτό είναι ο τίτλος. Ας ελπίσουμε για την ομάδα μου. Υπάρχει ένα πράγμα που έχει σημασία τις επόμενες εβδομάδες, αυτή τη νέα αρχή για την Ευρώπη εκτός από τη νέα διακυβέρνηση της Ευρωζώνης να φέρεται και αυτό που θέλουμε ε, μια ευρωπαϊκή πράξη για ε, ανάκαμψη και ε, οι Αμερικανοί το έχουν κάνει αυτό από το 2009. American Recovery and Stimulus Act. 800 δις ε, ε, στην υγεία, στις υποδομές, στην ενέργεια και φορολογικά κίνητρα ομοσπονδιακά για ε, μικρομεσαίες και για οικογένειες. Εμείς δεν το κάναμε και πέρασε το 8, το 9, το 10, το 11, το 12 και το 13. Και 2 με 3% ήταν εκτοτή ανάκαμψη, 2,2% στην Αμερική, για φέτος 2,2%. Και υπάρχει μια διαφορά εκεί. Γι' αυτό θέλω να υπογραμμίσω σε αυτή τη σημερινή συνεδρίαση αυτό είναι κάτι άλλο από το να ξαναβρεις κάποια άλλα δισεκατομμύρια και να τα πακετάρεις με άλλο τρόπο. Από λεφτά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή από άλλες γραμμές του προπολογισμού με αναδιατάξεις. Θέλουμε μια γνήσια τέτοια προσπάθεια και η ομάδα μου θα κάνει δικές της προτάσεις τις επόμενες ημέρες. Έχουμε χάσει μια δεκαετία. Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλη μία. Τώρα θα πρέπει να ναι. δράσουμε. Ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ, ο κύριος παρακαλώ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπε και ο Πρόεδρος, η πρόσφατη έκθεση εμπειρογνωμόνων για το κλίμα είναι άκρο σημαντική. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ανησυχητική φωνή που θα πρέπει να μας κάνει να επαγρυπνήσουμε και να δράσουμε κατεπηγόντως. Και βεβαίω το σημαντικότερο αποτέλεσμα το περιμένουμε στη Σύνοδο των Παρισίων το Δεκέμβριο του 2015. Αυτή η έκθεση των εμπειρογνωμόνων ε, δίνει στοιχεία πραγματικά ανησυχητικά, διότι προβλέπει ότι οι κλιματικές αλλαγές θα έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις που θα είναι και ιδιαίτερα εκτεταμένες και αμετάκλητες. Ε, ιδίως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα έχουν φτάσει ε, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και 800.000 χρόνια. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό το φως αυτών των ε, ε, ανησυχητικών σχολείων έλαβε κάποιες αποφάσεις. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω με αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, ότι μπορούμε να τις λάβουμε ως ένα σημείο αφετηρίας, γιατί φοβάμαι ότι θα έπρεπε να έχει γίνει μια επί της συζήτηση κάποιων στοιχείων που αυτή τη στιγμή υπόκεινται και υποκρύπτονται σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Εκεί φαντάζομαι ότι υπάρχει βασική διαφωνία μεταξύ μας. Αλλά η αρχή της ανταγωνιστικότητας, την οποία ακούω διαρκώς να επαναλαμβάνεται μόλις προηγουμένως σε πολλούς τομείς, όπως ο τομείς, ο τομέας των μεταφορών δεν συνάδει με τους στόχους που υποτίθεται ότι θέλουμε εδώ να επιτύχουμε. Το να συνεχίσουμε να ευνοούμε τα οχήματα, τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα εις βάρος των σιδηροδρόμων λόγου χάρη, αυτό δεν ε, εξυπηρετεί νομίζω τους στόχους μας εκτός από και άλλα θέματα, κινδύνους για το νερό ή την εκτατική, τις εκτατικές καλλιέργειες στον τομέα της ε, γεωργίας. Δηλαδή πλήττεται και το περιβάλλον και αντίκενται όλα αυτά και στους κλιματικούς μας στόχους. Θα πρέπει λοιπόν αλλιώς να ε, ακουστεί η φωνή μας, όχι μόνο ως προς τις ε, ευκαιρίες για οικονομικά κέρδη με το σχιστολιθικό αέριο ή τα, το πετρέλαιο ή άλλα ή την πετρελοφόρο άμμο και άλλα πράγματα που σκεφτόμαστε εδώ να εισάγουμε. Δεν ξέρω λοιπόν αν υπάρχουν λύσεις μακροπρόθεσμες εάν δεν παντρέψουμε ένα άλλο είδος οικονομικής ανάπτυξης το παραγωγικό μας μοντέλο να λάβουμε υπόψη περισσότερο την εξοικονόμηση ενέργειας και την λιγότερη ρήπανση και βεβαίως με εργαζομένους οι οποίοι να έχουν υψηλά προσόντα και να λαμβάνουν και τις κατάλληλε αμοιβέ. Ε, εδώ λοιπόν κύριε Γιούνκερ, ε, εάν έχετε ένα μεγάλο πρόγραμμα υποδομών να το στηρίξουμε. Έχετε κάτι τέτοιο τα αστικά κέντρα, τις μεταφορές, τη στέγαση, ε, τη ζωή της πόλης, διότι ταυτόχρονα και οι δημόσιες υπηρεσίες είναι ο καλύτερος ρυθμιστής όλων αυτών των αλλαγών και των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης από τη Σύνοδο της Κοπενχάγης υπήρξαν κάποιες οικονομικές δεσμεύσεις. Θα πρέπει να κάνουμε αρκετά γιατί και απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε κάποιες ε, υποχρεώσεις. Ξέρουμε πόσο θα δυσκολευτούν στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε το θέμα της επιδημίας του έμπολα. Ε, μεθαύριο θα έχουμε λόγω των κλιματικών αλλαγών και άλλα σοβαρότερα ε, ανθρωπιστικά προβλήματα από τους μετανάστες λόγω των κλιματικών αλλαγών. Στις συζητήσεις λοιπόν στο Συμβούλιο βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ε, το Συμβούλιο περισσότερο ε, συνάδουν προς το στόχο της μείωσης του 70% ε, μέχρι το 2050 για να περιοριστούμε στους δύο βαθμούς θερμοκρασίας μας. Λάμπερτς, καταρχήν ευχαριστώ τον κύριο Λεγιαρίκα ε, για αυτά που είπε, τα οποία και στερνίζομαι απόλυτα, δεν θα τα επαναλάβω. Υπάρχει το θέμα όπως βλέπουμε το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Για τους στόχους για το κλίμα. Αν ε, το θεωρήσω αισιόδοξα, λέω τουλάχιστον 40% των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα είναι περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στον πλανήτη. Άρα έχουμε ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν συγκρίνω τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο, διαπιστώνω ότι όντως είμαστε πιο αισιόδοξοι από τους άλλους εταίρους. Αν όμως ε, ε, λάβουμε υπόψη την επιτακτική ανάγκη που έχει ο πλανήτης να μειώσουμε τις εκπομπές αέριου του θερμοκηπίου, τότε βλέπω ότι στερούμε σχέση με τους στόχους. Λέμε τουλάχιστον 40% μπορεί να είναι περισσότερη η μείωση, αλλά δεσμευτικό σήμερα είναι ο στόχος του 40% και από οικολογική άποψη είναι ανεπαρκή στόχος για να υλοποιήσουμε ε, τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Φυσικά δεν μπορεί η Ευρώπη μόνη της να υλοποιήσει τους στόχους. Συλλογική και διαφοροποιημένη ευθύνη, λένε οι Κινέζοι. Όταν όμως γνωρίζουμε ε, ποια είναι η ευρωπαϊκή ευθύνη για το στόκ διεξουδίου του άνθρακα, θα έχουμε πραγματικά αυξημένε ευθύνες. Τώρα για τους άλλους δύο στόχους, 27%, ε, τα δύο ποσοστά 27%. Κανένας δεν είναι ε, δεσμευτικός από τους δύο στόχους του 27%. Ούτε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από τη στιγμή που δεν είναι δεσμευτικός ο στόχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς θα τον επιβάλλεται έχουμε δύο στόχους που είναι προαιρετικοί και άρα δεν θα υλοποιηθούν. Γνωρίζουμε ότι στο πακέτο των 20% τριών ποσοστό του 20% όσες υποχρεώσεις δεν είναι δεσμευτικές δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Αν δεν υπάρχουν μετρήσιμοι στόχοι και υποχρεωτικοί δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Έχουμε οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Από τη στιγμή που έχουμε, ε, οι φιλόδοξοι στόχοι σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν και οικονομικό και στρατηγικό χαρακτήρα. Θα πρέπει ως Ευρωπαίοι να ε, αποφασίσουμε ή θα πρωτοστατήσουμε σε αυτή τη βιομηχανική επανάσταση ή θα την εισαγάγουμε από τους ε, εταίρους μας. Γιατί αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να επιβραδύνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άρα θα μας προλάβουν και θα μας ξεπεράσουν οι εταίροι μας. Είναι και στρατηγικό αυτό ο στόχο, γιατί ποιοι τίποτα τα χέρια τη, οι προμηθευτέ ορυκτών καυσίμων στην Ευρώπη και κυρίω ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Άλλεν λέει, ε, αφήνει τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αφήνει την, ε, ε, την ενεργειακή απόδοση Ευρώπη να υστερεί. Εμεί θα υποφεληθούμε. Δύο σημαντικά λάθη και σε οικονομικό και στρατηγικό επίπεδο για τι κλιματικέ αλλαγέ και του στόχου μα. Στην πρώτη παραγράφο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, το Συμβούλιο επιφυλάσσεται να επανέλθει στις λεπτομέρειες του θέματος. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και μάλιστα ομόφωνα αποφασίζουν. Δεν είναι αυτή η νομοθετική διαδικασία που προβλέπει η συνθήκη. Επουδενή δεν πρόκειται να δεχτούμε αυτή την τρικλοποδιά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γιατί είμαστε συναρμόδιοι νομοθέτες. Δεν θα μας φέρει το Συμβούλιο πρωτοτελεσμένο γεγονότος επειδή ήταν δύσκολη η επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς αυτή την κατάσταση γιατί ελοχεύει εδώ κίνδυνος ε, μιας θεσμικής ε, τρικλοποδιάς. Ο κύριος Νάταλ εκ μέρους της ε, Άμεσης Δημοκρατίας και Ελευθερίας. Um, well... Κύριε Πρόεδρε, όλοι είναι πρόεδροι εδώ βέβαια. Πάντως βλέπουμε στον κύριο, τον κύριο Φάναρο που είναι στην τελευταία του διάσκεψη Προέδρων. Ε, τι θα πείτε για την Ουκρανία, την ενέργεια, την οικονομία. Ε, όλα αυτά που συζητήθηκαν νομίζω ήταν τα συνηθισμένα. Σας παρακολουθώ εδώ και πέντε χρόνια και ήθελα να κάνω και ένα επικριτικό σχόλιο για όσα άκουσα. Ε, τον περισσότερο καιρό μου θυμίζατε τον άλλο γνωστό πολιτικό του καιρού μας Ε, τον, κύριο Χάλι, ο οποίος ε, στα πλαίσια του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσέιν κατέληξε να είναι απλώς ένας γραφικός. Με συγχωρείτε, Μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή περιμένετε κύριε συνάδελφε. Μια στιγμή περιμένετε. Είχε ψευδεστήσεις και σε βαθμό που δεν είχε καμία συνέστηση. Αυτό βλέπω να σημαίνει εγώ και τα τελευταία πέντε. Εντάξει, μια στιγμή, περιμένετε, δεν γίνεται έτσι. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, περιμένετε. Δεν μπορείτε τον πρόεδρο ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να το συγκρίνετε με τον Υπουργό Προπαγάνδας μιας αιμοσταγούς δικτατορίας. Das ist deutlich. Είναι σαφέστατα περισσότερα. Μια, μια στιγμή, περιμένετε, συγκρατηθείτε λίγο είναι πολύ περισσότερο από την αντιπαράθεση και με συγκρούσει στην κοινοβουλευτική ε, δημοκρατία. Λοιπόν, σας εγκαλώ στην τάξη να αποφεύγετε τέτοιες εκφράσεις ή όσο είμαι εγώ πρόεδρος εδώ στο Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να υπολογίζετε τις εκκυρώσεις για να το καταλάβετε αυτό ξεκάθαρα. Παρακαλώ. Okay, I will carry on then. Εντάξει λοιπόν, θα συνεχίσω. Τι πετύχατε λοιπόν σε αυτή την πετέτεια ω ε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Καταστρέψατε τη δημοκρατία στην Ελλάδα και την Ιταλία, διότι τελικά δύο πρωθυπουργοί έχασαν ε, τη θέση του. Επιβάλατε ε, όλες αυτές, όλους αυτούς τους περιορισμούς από τις Βρυξέλλες. Διογκώθηκε η ανεργία των νέων με 50% στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Με τόσα εκατομμύρια πολίτες που ζουν σε συνθήκε απελπιστική φτώχεια δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Ε, στην ε, Ισπανία, ε, οι Ισπανοί μετασταναστεύουν στην Αργεντινή, οι Πορτογάλοι στην Βραζιλία. Και φαίνεται ότι όλοι οι υπόλοιποι έρχονται στη Βρετανία. Πέρυσι μόνοι μόνον είχαμε 275.000 μετανάστε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση από την υπόλοιπη, προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει οδηγήσει σε πτώση των μισθών και κάποιοι έχουν χάσει και τη δουλειά του. Όμω εσεί, κύριε Θαροποϊ Ακόμη ε, λέτε ότι θα πρέπει να ε, ε, νύπτετε τα σχήρα σας επιτρέποντας να ελέγχουμε μόνοι μας τα σύνορά μας. Εδώ πέρα λοιπόν τι θα γίνει και με την ε, επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς Ανατολάς, όταν όλοι δυτικά της Ουκρανίας πιστεύουμε ότι αυτό είναι μια καθαρή τρέλα. Είδαμε και τις εκλογές που οδήγησαν σε μια κατακαιρματισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε την κρίση της Ουκρανίας πέρσι. Βλέπουμε τώρα το φάσμα του αποπληθωρισμού να κρέμεται πάνω από όλα τα μεσογειακά κράτη. Νομίζω ότι η πενταετή σα θητεία ως, Ευρωπαϊκού, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Φαναρομπό, ήταν μια αποτυχία και βασίζεται στις ψευδεστήσεις, απελπισία και την ε, ε, πραγματική απογοήτευση. Τίποτε που θα πείτε σήμερα δεν θα μπορούσε να με κάνει να αλλάξω γνώμη. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μποριέτσι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν είχατε περάσει το πρωί σας μαζί με τους εργάτες που ήρθαν ε, από την Ιταλία, από τη σιδηρουργική βιομηχανία, θα ξέρατε γιατί θέλω να σταθώ σε κάποια ε, σημεία συγκεκριμένα. Εδώ Καλό θα ήταν να τα σκεφτείτε και εσείς κύριε Φαροποϊκέ, και για το παρελθόν σας ως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και για τους επόμενους ε, Προέδρους που θα μπορούσαν ενδεχομένως να να διορθώσουν κάποια ε, πράγματα, ακούγοντας όχι τους ε, διαξυφισμούς ε, που είναι λίγο ρητορική, επιδείξεις ρητορικής, αλλά τις αντιδράσεις εκατομμυρίων Ευρωπαίων ψηφοφόρων. Πώς τα σχολιάζετε ότι δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα, για να μην πω απολύτως τίποτα, για να μειωθεί η γραφειοκρατική οικοδόμηση της Ευρώπης, η οποία ακόμη και τώρα συνεχίζει να εφαρμόζει με το παράδειγμα που έδωσα μόλις τώρα ε, λανθασμένες επιλογές ως προς την ανταγωνιστικότητα. Η ανταγωνιστικότητα ε, σε ορισμένους τομείς είναι διεθνής. Οι παρεμβάσεις σας λοιπόν για να εμποδίσετε βιομηχανικές λύσεις που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την παραγωγή αριστείας στην Ευρώπη τελικά φρενάρονται. Ε, η αντικειμενική πραγματικότητα λέτε ότι είναι η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και τελικά χάνουμε το παιχνίδι λόγω των έξω ευρωπαϊκών παραγωγών αλλά για τα σημαντικά ζητήματα που συζητήθηκαν για τις εναλλακτικέ ε, πηγές ενέργειας, νομίζω ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε την εσφαλμένη πολιτική των κρατικών ενισχύσεων, ε, ε, αντί να έχουμε μια ελάφρυνση φορολογική για όλες τις χώρες με συγκεκριμένους στόχους. Εδώ θα πρέπει να στηρίξουμε τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά συγκεκριμένα, που δεν καταναλώνουν, που δεν πλήττουν την γη, την επικράτεια των ε, εδαφών ή να αξιοποιήσουμε τα απόβλητα των τροφίμων, να κάνουμε δηλαδή επιλογές εφής επιλογές που λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα και δεν τις ερμηνεύει μια ασφικτική γραφειοκρατία με τρόπο ε, κοντόφθαλμο. Δηλαδή θα πρέπει η Ευρώπη των, της παραγωγής, των εργατών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν να στηριχθεί. Μιλήσατε και για ένα μέσο που θα ενθαρρύνει την αντιδικοποίηση της παραγωγής, ε, βελτιώνοντας τη συμβολή στην παραγωγή με τα μέτρα καταπολέμησης της αποψήλωσης. Μα εδώ νομίζω η κοινή και η πολιτική έχει συμβάλει τα μάλα ήδη. Πώς ε, θα βελτιώσετε περισσότερο την περιορισμό των βασικών εκτάσεων με τις δημογραφικές αυτές τάσεις που υπάρχουν και με την απέτηση να αυξηθεί η παραγωγή. Βλέπουμε να λέγεται ότι η Ένωση πρέπει να εγγυηθεί ότι τα κράτη-μέλη δημιουργούν ένα σύνολο κινήτρων για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια που να είναι βιώσιμο και ε, σταθερό. Βάσει των προηγούμενων ενδείξεων. Να κλείσω λέγοντας ότι οι κατευθυντήριες ε, γραμμές για τις διαπραγματεύσεις TTIP ανατέθηκε η, εντο... η διαπραγματευτική εντολή από το Συμβούλιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμως. Όμως βλέπετε τις αντιδράσεις των παραγωγών τροφίμων ήδη. Αυτό δεν θα έχει αντίκτυπο στην ενεργειακή πολιτική και σε όλες μας τις υπόλοιπες πολιτικές. Δεν έχουμε ήδη εδώ μια περιοχή αριστείας αναντικατάστατη δεν θα πρέπει να τα υπερασπιστούμε με νύχια και με δόντια αν θέλουμε να υπερασπιστούμε την Ευρώπη των λαών και όχι την Ευρώπη των τραπεζιτών που τόσο πολύ βρίσκεται στην ε, ε, καρδιά των ε, θειασωτών της Bilderberg και του κτηρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Βίνκελ έχει τώρα πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Πέντε λεπτά έχω. Για να απαντήσω σε όλες τις ε, προτάσεις, ε, σε όλα τα επιχειρήματα. λίγο είναι ο χρόνος και θα αναφερθώ σύντομα στις παρεμβάσεις. Δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν πολλοί πρωθυπουργοί μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πάντα έχω την εντύπωση μετά από μια μακρά εμπειρία που έχω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπάρχει για να λύνει προβλήματα, όχι να τα ε, διευρύνει και να τα ενισχύει. Και ε, επί μακρόν σημείωνα και πάντα συνέκρινα τα όσα διαμείβονται εντός της και με τις δηλώσεις που γίνονται μετά. Και καμιά φορά δεν συνέπιπταν οι σημειώσεις μου με αυτά που άκουγα μετά. Πρέπει να πω στον καλό μου φίλο το Ματέο Ρέντζι ότι δεν είμαι πρόεδρος συμμορίας γραφειοκρατών. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι πολιτικό όργανο και όχι μόνο όργανο, αλλά και θεσμικό όργανο. Και καλό όλους τους πρωθυπουργούς να σέβονται αυτό το θεσμικό όργανο γιατί δεν έχουμε λιγότερη νομιμότητα από κάποιους άλλους. Αν είχα ακούσει, αν άκουγα ή ο κύριος Μπαρόζο μόνο τους γραφειοκράτες, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον προπολογισμό της Ιταλίας η Κομισιόν θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και δεν δέχομαι, δεν ανέχομαι αυτές τις επιπόλαιες κριτικές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αξίζει καλύτερη συμπεριφορά η Κομισιόν από αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Και αφού άκουσα και τον κύριο Καμάλ, πρέπει να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζετε εσείς τα πράγματα, λέγοντας ότι έτσι τα ε, βλέπει ο κόσμος, όχι, δεν ισχύει αυτό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα πράγματα, ε, όχι όπως τα βλέπει κανείς, η κοινή γνώμη στη Βρετανία. θα πρέπει να παρουσιάζονται με σεβασμό στους κανόνες των συνθήκων. Ερωτήσεις τώρα όχι. Δεν τέλειωσα. Θα έχετε και άλλες ερωτήσεις άμα τελειώσω. Περιμένετε. Θα ήθελα λοιπόν να πω ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού εφαρμόζει τους κανόνες όπως έχουν κατοχυρωθεί από τα κράτη-μέλη. Επειδή όμως υπάρχει πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν προσκλήσεως της Ιταλικής κυβέρνησης εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα λυθεί το πρόβλημα. Το φετινό πρόβλημα εφαρμόζοντας πάντα τους κανόνες και είναι μια τελείως διαφορετική διάσταση ε, σε σχέση με τα προηγούμενα που ζήσαμε, τα προηγούμενα χρόνια. Και η όλη διένεξη, ε, αν θέλετε να την πω έτσι, είναι 8-9 ε, δισεκατομμύρια, δηλαδή 250% επιπλέον από ένα άλλο ποσό που ήταν 3,5 δις. Λοιπόν, ψάχνουμε μια λύση, αλλά δεν θα το χαρακτηρίσουμε και ληστεία των Ευρωπαίων Γραφειοκρατών. Εφαρμόζουμε τους κανόνες που συμφώνησαν τα κράτη-μέλη. Και ε, καταρχήν θα προτιμούσα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τους ίδιους τους κανόνες. Τούτων λεχθέντων σκεφτόμαστε, προγραμματιζόμαστε για μια λύση ε, η οποία θα είναι λύση στο πρόβλημα. Ε, σωστή και όχι να βολεύει τον έναν ή τον άλλον. Και δεν αφορά μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και άλλα κρατημέλη. Ε, ο αντίκτυπος της εφαρμογής των μέτρων στον προπολογισμό είναι πολύ χειρότερος ας πούμε, για τις ε, κάτω χώρες παρά για το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι γενικότερο το πρόβλημα, δεν είναι βρετανικό. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Και θα ήθελα να τον στον Γκί Φερχόφστατ, ε, μιλάει για το πρόγραμμα της ε, ανάκαμψης. Ναι, θα πρέπει να κινητοποιούμε και καλύτερα τα κονδύλια που δεν απορροφώνται. Με σύνεση καλύτερα. Γιατί να τα αφήσουμε εκεί χωρίς απορρόφηση. Δεν είναι αυτή η βασική μου ιδέα βέβαια, αλλά όλοι οι μηχανισμοί παλιοί και νέοι που έχουμε στη διάθεσή μας και που θα έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα κινητοποιηθούν. Η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή και θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία της ε, ε, ανάπτυξης και της απασχόλησης. Και δεν θα μπω σε συγκρίσεις τώρα. την κατάσταση Ευρώπης-Αμερικής με έναν τρόπο άκοψο που το έκανε ο κύριος ε, Φερχόφστατ. Άλλη είναι εντολή της Federal Reserve και άλλη της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας. Και δεν είναι γεγονός ότι ούτε το 8, ούτε το 9, ούτε το 10 δεν αρχίσαμε προγράμματα. Το κάναμε. αλλά δεν θέλησαμε να αυξήσουμε τα ελλείμματα και τα χρέη. Δεν θέλουμε να μπούμε σε συγκυριακά λεγόμενα προγράμματα που δεν εξυπηρετούν τίποτα παρά μόνο να τρέφουν ψευδεστήσεις και ρίχνουν ε, πραγματικά ε, λάδι στη φωτιά και δεν βοηθούν στην Ευρώπη. Μου λέει ο φίλος ο Πιτέλα ότι είμαι συμπαθής. Εντάξει, αντικειμενικό αυτό δεν λέω αλλά πολύ αυστηρός λέει. Κοιτάξτε, ακούστε με. Ότι δείχνω λέει αυστηρός. Μα είμαι αυστηρός. Γιατί όταν μιλώ για την απασχόληση δεν έχω λόγο να χαίρομαι. Όταν είσαι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντιμετωπίζεις μια κατάσταση όπου πάνω από 25 εκατομμύρια είναι οι άνεργοι, όταν είσαι απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση οικονομική, ε, δεινή και επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, πώς να χαρεί κανείς, πώς να γελάσει. Πρέπει να είμαι αυστηρός, γιατί θέλω να είμαι αυστηρός με τον εαυτό μας. Εκείνοι που είναι ε, στην ανεργία, στη φτώχεια και αναξιοπαθούντες δεν γελάνε. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι σε όλα αυτά. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Merci Σας ευχαριστώ για τη δέσμευση και τις απαντήσεις και την προσήλωσή σας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο για πέντε λεπτά στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστώ για αυτό το πεντάλεπτο. Θα είναι το τελευταίο μου πεντάλεπτο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ποτέ δεν ξέρει κανείς. Όχι, ξέρει, ξέρει, σίγουρα, 100%. Ούτε θα ζητήσω πλέον πεντάλεπτο. Ούτε το ζήτησα εγώ προηγουμένως. Για τα θέματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το κλίμα και την οικονομική κατάσταση. Για το κλίμα. Ευχαριστώ όλους όσους ε, σχολίασαν το ζήτημα του κλίματος. Γιατί λέμε ότι η πολιτική ασχολείται μόνο με βραχυπρόθεσμα θέματα. Όχι, αυτή τη φορά ασχοληθήκαμε και με μακροπρόθεσμα. Το κλίμα είναι μακροπρόθεσμο θέμα. Και ευχαριστώ θερμά όλους όσους μπήκαν στον κόπο να αναπτύξουν τις ιδέες τους για τα θέματα του κλίματος. Δεν, δεν θα κάνουμε συναγωνισμό ποιος είναι πιο φιλόδοξος. Πάντα μπορούμε να είμαστε φιλόδοξοι ως προς τους στόχους μας. Το δικό μου πρόβλημα και το πρόβλημα του διαδόχου μου θα είναι να συνδυάσουμε τις φιλοδοξίες μας με την επίτευξη συμφωνίας από τις 28 χώρες μέλη. Και αυτός ο συνδυασμός είναι δύσκολος. Είμαστε φιλόδοξοι. Να σας δώσω δύο στοιχεία. Και θα τα υλοποιήσουμε. Ε, μείωση κατά 20% του διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με τις τιμές του 1990. 20% μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μέσα σε 30 χρόνια. Τώρα θέλουμε μείωση κατά 40%, επιπλέον 20% δηλαδή, μέσα σε 10 χρόνια. Αυτό είναι αρκετά φιλόδοξο στόχος. Και μάλιστα το καταφέραμε στην εσωτερική αγορά. Και το ζητάμε στην εσωτερική αγορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγέ διοξιδίου του άνθρακα με του παγκόσμιου εταίρου μα για να απαλλαγούμε από τι δικέ μα ευθύνε. Είπαμε εσωτερική προσπάθεια, εγχώρια προσπάθεια για τη μείωση αυτή. Ως προς τη φιλοδοξία λοιπόν νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξη η συμφωνία. Θα πρέπει φυσικά να λάβουμε υπόψη τις ετερότητες και τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Φανταστείτε να μην είχαμε καταλήξει συμφωνία. Σε τι θέση θα ήμουνα εδώ σήμερα. Θα φαινόταν ότι η Ευρώπη υστερεί, ότι δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Και θα μας έλεγε και ο Γενικός Γραμματέας ότι η Ευρώπη δεν ανταπεξήλθε στις προσδοκίες που είχε γύρει. Και γι' αυτό και προσπαθούσαμε τους τελευταίους δύο μήνες, όχι σε, μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε όλε τι προπαρασκευαστικές δράσει, για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Στηριχθήκαμε στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ω προ τους τρει στόχους και το βαθμό δεσμευτικότητάς τους. Βασιστήκαμε στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως διαμορφώθηκαν πριν από μερικούς μήνες. Και ο στόχος για τη μείωση κατά 40% είναι ο κύριος στόχος, ο κεντρικός στόχος. Γιατί για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο θα πρέπει να επενδύσουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα πρέπει να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Αν δεν το κάνουμε, δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε τον φιλόδοξο στόχο τη μείωση κατά 40% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και για τι οικονομίε στην ενέργεια, για την εξοικονόμηση στην ενέργεια, ούτε στην προηγούμενη φάση είχαμε υποχρεωτικού χαρακτήρε. Ήταν προαιρετική, ενδεικτική η στόχη, δεν ήταν δεσμευτική. Θα πρέπει λοιπόν να συμφιλιώσουμε, να συνδυάσουμε τι φιλοδοξίε μα με τον απαραίτητο ρεαλισμό. Και πιστεύω ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και αν θέλουμε να τελειώσουμε με ένα αισιόδοξο τόνο. Νομίζω ότι αυτό τον αισιόδοξο τόνο δίνει η φιλόδοξη αυτή συμφωνία για το κλίμα. Φυσικά μπορούμε να είμαστε πιο απαιτητικοί, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και μπείτε στη θέση μου λίγο. Έπρεπε να βρούμε συμφωνία που να τη δεχτούν και 28 χώρες μέλη. Και σας διαβεβαιώ ότι υπήρχαν σημαντικές αποκλήσεις, διαφωνίες και αυτό είναι εφημισμό η χρήση Τώρα, για την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει ε, πανάκια για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να γίνει ανάλυση και προσπαθήσαμε να κάνουμε μια τέτοια ανάλυση και μάλιστα εμπεριστατωμένη της κατάστασης με απότερο στόχο το να δημιουργήσουμε θέσει απασχόλησης και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη. Αλλά η κατάσταση είναι περίπλοκη γιατί για την νομισματική πολιτική Ήδη έχουμε μια ευνοϊκή πολιτική, όπως λένε πολύ, αλλά και για τη δημοσιονομική πολιτική και η πρόσφατη σημερινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το επιβεβαιώνει και για τη δημοσιονομική πολιτική έχουμε ουδετερότητα του αποτελέσματος στην οικονομία για το 2014 και το 2015. Ουδετερότητα. Δηλαδή, η δημοσιονομική πολιτική δεν είναι η αιτία της ε, μικρής οικονομικής ανάπτυξης. Ούτε σε αυτήν ε, οφείλεται η ύφεση. Και μπορείτε να ελέξετε τα στοιχεία που σας δίνω. Κανείς φυσικά δεν ζητάει μια πολιτική deficit spending. Κανένας δεν υπέρ μιας τέτοιας πολιτικής. Γιατί γνωρίζουμε πού θα μας οδηγούσε μια τέτοια πολιτική. Για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μιλήσαμε. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο την ενιαία αγορά, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, στον ψηφιακό τομέα και στην καινοτομία και είμαι βέβαιος ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Γιατί εκεί χρειαζόμαστε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και θα πρέπει φυσικά να τονώσουμε και να αναζωπυρώσουμε τις επενδύσεις. Γιατί οι επενδύσεις υστερούν ε, σε σχέση με το επίπεδο επενδύσεων που είχαμε πριν από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση σε όλες τις χώρες. Ακόμη και τις χώρες που έχουν τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις. Και εκεί το επίπεδο επενδύσεων είναι χαμηλότερο από το επίπεδο επενδύσεων που είχαμε πριν από μία επταετία ή οκταετία. Γιατί, μεταξύ άλλων, γιατί και το χρέος των οικοκυριών, το ιδιωτικό χρέος είναι υπέρογκο και το ιδιωτικό χρέος δημιουργήθηκε κατά την πρώτη περίοδο της ιστορίας του ευρώ. Και αν μιλάμε για χαμένη δεκαετία, η πρώτη περίοδος Ευρωζώνης χαρακτηρίστηκε από σημαντικά λάθη. Αυτά τα λάθη ε, εμποδίζουν την ε, τόνωση των επενδύσεων. Γιατί αν δεν είχαμε ε, τόσο υψηλή ιδιωτική χρέωση, δεν θα είχαμε τέτοια αποθάριση των επενδύσεων. Γι' αυτό και είναι σημαντικές και ευληματικές οι πρωτοβουλίες για τις επενδύσεις που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναζωπηρώσει και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Φυσικά έχουμε κάποιες συλλογικέ ανάγκες, αλλά και το θέμα των ιδιωτικών επενδύσεων έχει κέρια σημασία και θα βρεθεί στο επίκεντρο των μελλοντικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε πολλά μέσα στη διάθεσή μας, θα πρέπει όμως να προηγηθεί μια διεξοδική ανάλυση του παρελθόντος και της κατάστασης Ευρωσόνης. Ο Γκίφερ Χόφστατ ε, έκανε ένα παραλληλισμό με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Φανταστείτε να μην είχαν το σχιστολιθικό αέριο ή το σχιστολιθικό πετρέλαιο οι Αμερικανοί. Τότε θα είχαν ε, ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης παρόμοιους με τους δικούς μας. Δεν λέω ότι δεν ενήργησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε πιο έξυπνα σε ορισμένου τομεί από εμά. Στον τραπεζικό τομέα, για παράδειγμα, έβαλαν μία τάξη πολύ πιο νωρίς από μας. Ενεργοποιήθηκαν πολύ νωρίτερα. Εμείς ε, την, περασμένη, ε, την προηγούμενη Κυριακή δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα για τα τεστ κοπόσεως των τραπεζών. Αυτά τα τεστ ήταν απαραίτητα για να ξαναδημιουργηθεί ρευστότητα, που είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάκαμψη και για την τόνωση των επενδύσεων. Φυσικά μπορεί να διδαχθούμε από τους άλλους και Κάναμε και εμείς λάθη, αλλά πολλές φορές πληρώσαμε λάθη του παρελθόντος. Και εν κατακλείδη θα ήθελα να πω κάτι που δεν έχω κάνει συχνά, να μιλήσω στα Ολλανδικά. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα επαφές και με τους πρόεδρους των πολιτικών ομάδων, με μεμονωμένα μέλη δεν είμαι υπόλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό το λένε ξεκάθαρα οι συνθήκες, αλλά μέσω άτυπων επαφών, επαναλαμβάνω, άτυπων επαφών, έκανα πάντα ε, μια προσπάθεια ε, να ε, σας ενημερώνω. Μπορεί να διαφωνούσαμε και το παράδοξο τη συνθήκη τη Λισαβόνα ποιο είναι. Δημιούργησαν τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρί οργανικού δεσμού όμω ε, ή σχεδόν καθόλου με τα θεσμικά όργανα. Α πούμε, τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδόν καμία σχέση. Ουδεμία με το ευρώ και την ευρωζώνη, σχεδόν καμία ε, με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, εκτός από την ενημέρωση αυτή. Οπότε αυτό που δεν υπήρχε τυπικά έπρεπε να δημιουργηθεί άτυπα. Και γι' αυτό προσπάθησα να το πράξω κι εγώ ε, στο βαθμό που τα θεσμικά όργανα ως όργανα ε, θα πρέπει να εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν ήταν εύκολο εγχείρημα πάντα, αλλά τα καταφέραμε. Όταν ε, έπαιρνε πρωτοβουλίες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την νομοθετική διαδικασία και για το κλίμα θα ακολουθήσει τώρα, όποτε υπήρχε νομοθετική διαδικασία και τελικά συμφωνούσαμε, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ε, πρωθυπουργοί που είναι επικριτικοί προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάντα εγώ σας υπερασπιζόμουν ότι ε, άμα πας στο Κοινοβούλιο νομίζω ότι είναι όλοι στην αντιπολίτευση γιατί είναι πολύ επικριτικοί αλλά τελικά καταλήγουμε πάντα κάπου και στο δύσκολο εγχείρημα και στην άσκηση ε, του προπολογισμού. και για μένα αναφέρω 28 στην ίδια γραμμή και μετά σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι υπηρετούμε την ίδια υπόθεση, την, την ευρωπαϊκή υπόθεση. Και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα τελευταία πέντε έτη προσπάθησαν όσο γίνεται να συνεργάζονται και ε, να ήταν το πιθανότερο ε, η πιο δύσκολη περίοδος που έζησε η Ένωση ε, από τη δημιουργία της. Το είπα και προηγουμένως. Το θέμα ε, είναι ότι ε, τα προβλήματα, ε, ορισμένα από αυτά τα είδαμε μόνο ακροθυγώς. Στην επόμενη πενταετία θα πρέπει να αποδείξουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη και η επιστροφή της εργασίας είναι δυνατή. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα είναι πολύ διαφορετική, δυστυχώς και πολύ πιο αρνητική η έκβαση των επόμενων ευρωεκλογών. Τα επόμενα πέντε έτη θα είναι ακόμα πιο σημαντικά πολιτικά από ό,τι τα προηγούμενα. Σας ευχαριστώ και πάλι για όλη τη συνεργασία που είχαμε. Adieu, au revoir. Στο επανειδήν. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, για τα λόγια σας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για το μήνυμά σας αυτό προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσουμε και θέλουμε να διαδραματίσουμε κι εμείς ένα σημαντικό ρόλο στην ερχόμενη πενταετία, συμβαδίζοντας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χέρι-χέρι, για να δώσουμε τις απαντήσεις που χρειάζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτή την πρόκληση έχουμε μπροστά μας και θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τα λόγια σας, τη δουλειά σας και το, ε, τα λόγια εμπιστοσύνη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που υπερασπιστήκατε και την πολυγλωσία και μιλήσατε για τη μετρική σας γλώσσα. Η πολυγλωσία είναι ε, κάτι το ζωτικό για το Ευρωκοινοβούλιο. Και τώρα ο κύριος Μποργέτσιου που δεν είναι εδώ, οπότε ευθύς αμέσως ο λόγος στον κύριο Νούταλ. Κύριε Πρόεδρε, σε μια από τι τελευταίε σα κινήσει ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Φαρόπα, και με τη βοήθεια του κυρίου Μπαρόζο, ουσιαστικά οδηγήσατε σε ενέδρα τον ε, Βρετανό Πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με το 1,7 δι στελίνε. και τώρα η κυβέρνησή μα θα πρέπει να επιβαρύνει του Βρετανού προλογουμένου για να πληρώσουν αυτό το λογαριασμό. Διότι δεν πετύχαμε ακριβώς το... γιατί πετύχαμε ακριβώς το στόχο μας και από ό,τι φαίνεται η επιτυχία τιμωρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κάμερον είπε ότι δεν θα παραχωρήσει αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι αλλά παρόλα αυτά εσείς είπατε ότι θα επιβληθεί πρόστιμο αν δεν ε, καλύψουμε αυτή την υποχρέωση. Να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον κύριο Φαρόμπο και τον κύριο Μπαρόζο, διότι ε, πετύχατε την Βρετανία προς την έξοδο τελικά και νομίζω ότι αυτό θα υλοποιηθεί και ελπίζω ότι αυτό θα υλοποιηθεί πολύ σύντομα. Κύριε Λάμπερτ, έχετε το λόγο. Κύριε Φαρομπόη, όταν ε, διοριστήκατε, ήμουν από αυτούς που σας υπερασπιστήκατε λέγαν κάποιοι, ένας πολιτικός από μια μικρή χώρα, χωρίς σοβαρό κύρος, ο Τόνι Μπλερ ήταν ο μεγάλος ηγέτης που θα έπρεπε να βγάλει από τον οικονομικό μερασμό την Ευρώπη. Εγώ είχα απαντήσει σε αυτούς τους ανθρώπους ότι θα σας εκπλήξει ο κύριος Φανοπόη. Και το καταφέρατε. Βέβαια, ε, εγώ σας γνώριζα, αλλά τελικά δεν εξεπλάγει τόσο όσο θα ήθελα. Διότι υπογραμμίσατε στην παρέμβασή σα ότι τελικώ η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Το είπατε για το κλίμα. Ε, ένα θέμα ήταν το να είμαστε φιλόδοξοι για να μην υπάρξει συμφωνία και άλλο ήταν να καταλήξουμε όντω σε συμφωνία χειροπιαστή. Που είναι, αν και μετριοπαθή, έστω υπαρκτή. Ε, σας κατανοώ, αλλά να σα θέσω και το εξή ερώτημα. Όταν κοιτάζετε την κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και δεν θέλω να σα δείξω με το δάκτυλο απαραίτητο, θα απευθύνω το ερώτημα σε όλους μας. Ε, εάν η πολιτική είναι τέχνη του εφικτού, η αύξηση ετησίως κατά 1% του αριθμού των Ευρωπαίων που βρίσκονται σε συνδίκες του κοινωνικού αποκλεισμού και ε, φτώχειας, 27 εκατομμύρια Ευρωπαίοι σε ανεργία, ε, το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια όλες τις κρίσεις 1% των Ευρωπαίων πολιτών πλούτησαν από όλα αυτά. Τελικά ήταν η καλύτερη ιδέα η τέχνη του εφικτού να μας πετύχει αυτά τα αποτελέσματα, ήταν αυτά τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Νομίζω λοιπόν ότι εάν δούμε και κρίνουμε το αποτελέσματο μπορούσαμε να τα έχουμε πάει καλύτερα. Όπως είπα στον κ. Μπαρόζο πριν από δύο εβδομάδες, δεν ήσασταν ο μόνος υπεύθυνο, αλλά είσαστε μέρος της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το διάστημα. Και θα ήθελα από πλευρά σας τουλάχιστον να δίνετε λίγη περισσότερη έμφαση στο θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Διότι έρχεστε από την οικογένεια των χριστιανοδημοκρατών στην Ευρώπη και μιλήσατε για οικονομική ορθόδοξη προσέγγιση, αλλά για την κοινωνική δικαιοσύνη δεν πολύ μιλήσατε και αυτό πραγματικά με λυπεί. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λιγαρίκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις που δώσατε και για το έργο όλο του Διάστε με αυτό. Αλλά τώρα, κύριε Γιούγκερ μας είπατε ότι θα προεδρεύσετε στην ομάδα των τεσσάρων προέδρων για την Ευρωζώνη, αν κατάλαβα καλά. Από την άλλη, εσείς κύριε Βανρομπέ, μας είπατε μόλις ότι ε, υπάρχουν κάποιες εντολές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την εφαρμογή των κριτηρίων του Μαστρίχ των λεγόμενων. Ισχύουν όλα αυτά, αλλά όταν μια χώρα δεν σέβεται τα κριτήρια της συνθήκης του Μαστρίχτ δεν σημαίνει ότι δεν κάνει αντιμεταρρυθμίσεις όπως τις έχω χαρακτηρίσει και ε, ε, λιτότητα. Και αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε μεγάλη εμπλοκή και οδηγεί και στην ανεργία και στα υπόλοιπα προβλήματα που γνωρίζουμε. Ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εντάξει, έχει κάνει κάποιες αλλαγές σε σχέση με αυτό που γνωρίζαμε με τις παρεμβάσεις αλλά άλλο είναι να δίνεις ε, χαμηλά δάνεια σε τράπεζες, χαμηλότοκα και άλλο είναι να επιτρέπεις την πραγματική οικονομία να λειτουργεί. Και εκεί υπάρχει όντως εμπλοκή. Ε, ε, σωστά μιλήσετε για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αλλά αυτό οφείλεται σε ε, πολύ στα τεράστια τραπεζικά έξοδα με μερίσματα για μεγάλους ομίλους και οι μικροί και οι μεσαίοι δεν έχουν πρόσβαση στην δανειοδότηση από τις τράπεζες. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε αυτά τα θέματα σε αρκετό βάθος. Ο κύριος Φερχόφστατ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς κύριε Φανρόμποη, πιστεύω ότι κάνατε καλά τη δουλειά σας. Βέλγος πολιτικός. Ε. ο Βέλγος πάντα είναι στη γραμμή της καλής ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα γνωρίζουμε αυτά, τι σημαίνει αυτό. Και στο Λουξεμβούργο έχουν κάποια ιδέα, αλλά λιγότεροι από μας. Θα ήθελα όμως να μιλήσω για το εξής. Αυτό που δεν κατανοώ όλες τις επικρίσεις που ακούσαμε ότι δεν πάει καλά η Ένωση. Ναι, το ξέρουμε. Και η ανεργία και η οικονομική ανάπτυξη είναι χαμηλή. Έχουμε προβλήματα στις τράπεζες, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι όλοι αυτοί που λένε ότι ε, θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω, να έχουμε λιγότερη Ευρώπη. Ενώ το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι δεν έχουμε αρκετή ολοκλήρωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μια μικρή εταιρεία νέα που μπαίνει στο διαδίκτυο και βρίσκει μια καινούργια εφαρμογή. Στην Ευρώπη χρειάζεται 28 άδειε. 200 συμφωνίες πρέπει να κάνει με τηλεφωνικές εταιρείε κινητή τηλεφωνία πριν βγάλει την εφαρμογή σε όλη την Ένωση. Στη ΣΥΠΑ μία είναι η άδεια, τρει συμφωνίες με τρει εταιρείε κινητή τηλεφωνίας. Τα ίδια για τη χρηματοδότηση μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις εγγύσεις που υπάρχουν στην Αμερική. Ε, σε εμάς δεν μπορούμε. Έχουμε άλλο κολάτερα σε μια χώρα, άλλο σε άλλη. Λοιπόν, εγώ αυτό ζητάω, Ζαν Κλοντ, να είσαι φιλόδοξος ε, τα επόμενα χρόνια. Διότι αυτό μας διαφοροποιεί τα τελευταία χρόνια από τα άλλα μέρη του κόσμου. Η έλλειψη φιλοδοξίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέγκερ ich bin hier noch neu. Κύριε Φαν Rompuy, ε, είμαι νέος ε, και ε, βουλευτής και δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω ως βουλευτής αλλά ως πολίτης. Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για το περιβάλλον και για την ενέργεια. αυτά που ακούστηκαν για το Ηνωμένο Βασίλειο με προβλημάτισαν. Είπατε σωστά ότι θα πρέπει να τηρούμε τους κανόνες αλλά αυτά να τα ακούμε από ανθρώπους που δεν τήρησαν κατ' εξοχή τους κανόνες στη διάσωση του ευρώ, μου φαίνονται λίγο περίεργα και λίγο κομικά, διότι όλες οι υποσχέσεις που δόθηκαν όταν ήρθε το ευρώ έχουν αθετηθεί όλες. Και εγώ θυμάμαι την υπόσχεση για την απαγόρευση ε, οικονομικής βοήθειας και διάσωσης. Αυτό όμως που με θλίβει ιδιαίτερα είναι αυτά που ακούστηκαν για τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί αν σκεφτεί κανείς τι ενοχλεί τους Βρετανούς, βέβαια άκουσα και αυτά τα απαράδεκτα του κυρίου Νότελ, αυτό που τους ενοχλεί είναι ότι η Κομισιόν για να σώσει το ευρώ αργά αλλά σταθερά θυσιάζει την αρχή της επικορικότητας και συγκεντρώνει. Για να σώσει το ευρώ η Κομισιόν έχει ε, καταργήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών και τον εναρμονίζει. Και για να σωθεί το ευρώ, η αρχή ότι κάθε χώρα θα πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες για το χρέος της και για τις τράπεζές της και πάλι καταργείται και ε, το χρέος και τα ρίσκα των τραπεζών κοινωνικοποιούνται. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε, θα πρέπει να φροντίσουμε η Μεγάλη Βρετανία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ίσως ε, μπορώ να σας θυμίσω ότι παρά ε, αυτή την αντιπαράθεση παραμένει ο δεύτερος συνεισφορέας στην Ευρώπη. Για πείτε μας, για μαντέψτε κύριε Βέμπερ, ποιος θα πληρώσει όταν φύγουν οι ε, Βρετανοί. Κυρία Βαμπρέμπτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, είναι η πρώτη τελευταία σας παρουσίαση και θα τα πω με χαρά στην κοινή μας μετρική γλώσσα. Ε, με ανησυχεί πολύ η υπόθεση του κλίματος. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για πράγματα ε, που κανονικά είναι στο περιθώριο της ευρωπαϊκής υπόθεσης. Η τελευταία έκθεση IPCC για την κλιματική αλλαγή, θα τα πω σύντομα, έχει καταλήξει σε δύο πολιτικά συμπεράσματα. Πρώτον, είναι πολύ προφανές και το ξέρουμε από παλιά, αλλά θα το ξαναπώ. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός, είναι κυρίως ανθρωπογενής και μας απειλεί με δραματικές συνέπειες. Και δεν είναι 12 παρα 5, είναι 12 και 5. Δεύτερο συμπέρασμα, οι επιστήμονες έχουν κάνει τη δουλειά τους ξανά, ξανά, ξανά και ξανά. Υπάρχει επιστημονική δουλειά. Και τώρα καλούνται οι πολιτικοί να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε και να δούμε υπό το φως όλων αυτών τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το κλίμα και την ενέργεια. Τα επαναλαμβάνω και τα υποστηρίζω. Πολλά υπόθηκαν. Βεβαίως υπάρχει συμφωνία και αυτό είναι καλό νέο. Είδα και τα εγγόνια σας ωραία στη φωτογραφία, αλλά είναι δύσκολο θα ήταν δύσκολο να τα κοιτάξετε και εσείς τα μάτια και εμείς τα παιδιά μας αν δεν υπήρχε συμφωνία. Κλίμα. Διάσκεψη των Παρισίων. Μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον υπάρχει συμφωνία. Καλά, μην περιμένετε τώρα να ενθουσιαστούμε και να σας χειροκροτήσουμε η ομάδα μας. Υποστηρίζουμε μεν τη συμφωνία να είναι πολύ λίγο φιλόδοξη και θα προσπαθήσουμε παντού τους επόμενους μήνες να ε, την ενισχύσουμε, να την οξύνουμε και ώψη των Παρισίων, όπου ξέρετε έχει λόγο και το Κοινοβούλιο. Για τους στόχους πρώτα απ' όλα. Εμένα δεν με ανησυχεί πάρα πολύ πάντα το ποσοστό ή το ύψος, αλλά ε, το θέμα είναι να μπορούν να εφαρμόζουν τη στόχη Enforceable το λένε αυτό στα αγγλικά. Ε, στην ενεργειακή απόδοση. Και στο παρελθόν δεν είχαμε δεσμευτικούς στόχους, αλλά υπάρχουν τα αποτελέσματα. Ήδη τα βλέπουμε μπροστά μας στην Ευρώπη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν έχουμε ποντάρει στην ενεργειακή απόδοση. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα ε, σε όλες τις χώρες παρόλο που όλοι οι ειδικοί λένε για την ενέργεια, για το κλίμα, για τη φθηνή ενέργεια είναι όλα θέματα που είναι αλληλένδετα και χρειάζεται ενεργειακή απόδοση. Και, επίσης υπάρχουν παραθυράκια στη συμφωνία και θέλει προσοχή να μην δίνεται επιταγή λευκό και να υπάρχει δυνατότητα να παραμείνουμε και να επενδύουμε λέει και σε ορυκτά καύσιμα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει συμφωνία και αγαπητέ Χέρμαν σε εσά πιστώνεται αυτό. Αν δεν υπήρχε η δική σας προσπάθεια και η ομάδα σας και το επιτελείο σας δεν θα υπήρχε συμφωνία και θέλω να σας ευχαριστήσω και ολόκληρη ομάδα μου για όλη τη δουλειά που κάνατε τα τελευταία χρόνια. Και έχετε αποδείξει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα δεν είναι ο συσχετισμός των δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα τον επιθυμούσα διαφορετικό, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα, και τελειώνω, και θα πρέπει να το σκεφτούμε, είναι ότι κάθε φορά που πάνε οι πρωθυπουργοί στο Συμβούλιο σκέφτονται μόνο την ίδια τους την κοινή γνώμη στη χώρα τους θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ στο Κοινοβούλιο για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και πάλι ευχαριστώ, Χέρμαν. Thank you very much. Ευχαριστούμε ομιλητής, ο κύριος Βέμπερ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Δεν ήθελα να σχολιάσω τους συναδέλφους από το EFTT, αλλά όταν ακούω τους συναδέλφους του UKIP, τι θα κάνουν όταν βγουν, όταν δεν θα έχουν αυτό το κάλαθο αχρήστων που λέγεται Ευρώπη και μπορούν να πετάνε όλα στα σκουπίδια. Τι θα απογίνουν χωρί βαρβάρους αυτοί οι άνθρωποι όταν φύγουν από την Ένωση. Αυτά για τους λαϊκιστές. Και για το αν τηρούμε τους κανόνες που είπε ο κύριο Νούτελ και τι κάνουμε, ο κύριο Χένκελ συγγνώμη, δεν αποφασίζουν τα πολιτικά κόμματα, ευτυχώς αν τηρούνται οι κανόνες κύριε Χένκελ στο πολιτικό μας σύστημα, αλλά οι δικαστές. Δουλειά τους είναι και καλά κάνουν και το αποφασίζουν αυτοί. Και θέλω να πω και στον κύριο Κεμάλ και να το σκεφτεί, ότι στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να σου έρχεται η λυπητερή, το καταλαβαίνω. Και εγώ θέλω να παραμείνει η Βρετανία, αλλά αν αρχίσουμε να χαλαρώνουμε, ε, να μην πληρώνουν τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις κάποιες χώρες, θα τις πληρώνουν κάποιοι άλλοι. Και πώς θα το εξήγησε το κόμμα σας κύριε Χένκελ στη Γερμανία, ότι αν ενδώσουμε στους Άγγλους θα τα πληρώσουν Γερμανία, Αυστριακή και λοιπή. Βεβαίως είμαστε υπέρ της στήριξης των κανόνων, αλλά να ισχύει για όλους όσοι εργάζονται εκεί. Και τέλος απευθύνουμε στο Χέρμαν Φαρόμποε τον προβόκαρα λίγο για να μας πει λίγο τα εσωτερικά του Συμβουλίου. Μας είπε ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα παραμείνει πιστός το ύφο του. Δυστυχώς δεν υπέπεσε σε αυτό τον πειρασμό. Δεν έμαθα τα εσωτερικά του Συμβουλίου. Δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ για το έργο και την εργασία σας και ό,τι επιθυμείτε για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Δεν είναι συζήτηση κύριε Κάμπον. Είναι διάσκεψη των Προέδρων. Ναι. Α, μπορείτε να δώσετε το λόγο σε κάποιον που δεν θα σας πλέξει το εγκόμιο. Διακόπτεται το μικρόφωνο. Λύεται η συνεδρία της διάσκεψης των Προέδρων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Βανερόμπο και τον Ζακ Κλόντ για την παρουσία τους. Θα πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες, κύριε Βουλευτά. Εντάξει, σαφές. Χαίρετε. Δύο φορέ ήδη μίλησε ο εκπρόσωπό σα. Ολοκληρώνεται η διάσκεψη των Πρόεδρων.